Good um, Καλημέρα σας. Είναι ένα δραματικό πρωινό με τις εκλογές στις Ηνωμένε Πολιτείε και σχεδόν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα των εκλογών. Φαντάζομαι ότι έχουν καθυστερήσει πολλοί συνάδελφοι λόγω του ότι παρακολουθούν τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Και εγώ σηκώθηκα πάρα πολύ νωρί και παρακολούθησα εκ του Μπορεί να έχουμε αποκλίνουσες απόψεις, σας μην το συζητήσουμε τώρα, αλλά όπως το έθεσε ο Πρόεδρος Ομπάμα, και ο ήλιος θα βγει και αύριο, ή, ε, όπως ο Λέναρτ Κοέν το είπε, για το καλοκαίρι, αλλά συνεχίζει τη ζωή. Ας περάσουμε τώρα στις εργασίες μας και συγκεντρωθούμε στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη. Καταρχήν την έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης, σας παρακαλώ. Δώστε προσοχή στο γεγονό ότι το σημείο 15 για τη διερευνητική αποστολή στα τέρατα ακυρώνεται λόγω τη ακύρωση ε, της επίσκεψης. Η εξήγηση είναι ότι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν μέλη του Κοινοβουλίου, δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση. Τώρα, η αίτηση 437 έχει προσθεθεί στο σημείο 26 σε ό,τι αφορά θέματα παιδικής πρόνοιας στη Γερμανία και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα υφετήσουμε την ημερησία διάταξη. Δεν έχουμε πρακτικά προσέγγιση και έχω τώρα κάποιες ανακοινώσεις. Θα σας χαίρομαι που σας ανακοινώσω ότι ένα μέλος του προσωπικού από το γραφείο του Ευρωπαϊκού Δημοσιολογητή, ο κυρίος Φιλίπ Κάιμοβιτς, ελπίζω να προφέρω το όνομά σας, κάπως αξιοπρεπώς, ε, μας επισκέπτεται στα πλαίσια μιας επίσκεψης μελέτης τρίμηνης στη Γραμματεία Πέτη για να ανταλλάξει απόψεις ε, και διδάγματα και να μας φέρει και τις δικές του εμπειρίες για το πώς ε, δουλεύει το γραφείο του Διαμεσολαβήτη και φυσικά να διαβάσει πώ λειτουργεί η δική μα γραμματεία στη δική του υπηρεσία. Το καλωσορίζω λοιπόν ένθερμα στην ομάδα και επίση ε, θεωρώ την ε, επίσκεψη μελέτη σα εδώ ω έκφραση τη πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ελπίζω λοιπόν ότι μία μέρα θα έχουμε και κάποιον από το δικό μας προσωπικό να επισκεφτεί το δικό σας γραφείο. Και πάλι καλώς ήλθατε. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το France Trua, που είναι εθνικό κανάλι τηλεόρασης, ε, αύριο θα ε, ένα τμήμα της συνεδρίασης ε, από τις 11. Και ουσιαστικά αυτό πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενημερωτικό σημείο. Όπως ε, Ξέρετε, όλες οι συνεδριάσεις μας ε, είναι να μεταδίδονται από το διαδίκτυο και αυτό εντάσσεται στην ίδια πρωτοβουλία. Να περάσουμε τώρα στο workshop, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες όπως παρουσιάζονται από τις αναφορές που λαμβάνει αυτή η Επιτροπή. Οργανώνεται από το θεματικό τμήμα ΓΑΜΑ και αυτό το θεματικό τμήμα εκπροσωπείτε σήμερα από τον Κλαβία Μαρζόκη. Σας καλωσορίζω, κύριε Μαρζόκη, εδώ στο βήμα. Επίσης, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω όσους είναι παρόντες σε αυτή την αίθουσα και όσους μας παρακολουθείτε από το σπίτι, από το διαδίκτυο. Όσοι παρακολουθείτε λοιπόν την ημερίδα δικαιωμάτων ανθρώπων με αναπηρία, όπω παρουσιάζονται από τι αναφορέ. Έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο γιατί έχουμε λάβει πάρα πολλέ αναφορέ που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Αρχικά, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες με εξαίρεση των τσοχικών, των εστονικών, φιλανδικών, λιθωνικών, πορτογαλικών και σλοβενικών. Η έχουμε και διερμηνία στην διεθνή νοηματική γλώσσα. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι έχουμε αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου και αυτό σημαίνει ότι θα καταγράφονται και οι παρεμβάσεις των ομιλητών. Όπως σας ανέφερα, αυτή η εκδήλωση ανήκει σε ένα κύκλο ετήσιων εκδηλώσεων που οργανώνει η Επιτροπή Αναφορών σε σχέση με τον ρόλο προστασίας που υλοποιούμε, του διαδραματίζουμε στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Όπως ξέρουμε, η σύμβαση είναι η πρώτη σύμβαση του ΟΗΕ που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα αναπηρίας και η πρώτη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνέφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Η σύμβαση διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους σε ίση βάση με τους υπολείπους. Πέρσι, Είχαμε μια ιστορική στιγμή στον τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την παρουσίαση της πρώτης έκθεσης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ενώπιον της Επιτροπής CRPD στη Γενέβη. Η Επιτροπή κατέληξε σε πάρα πολύ σημαντικές παρατηρήσεις ε, που άρχισαν εκείνη τη στιγμή να εφαρμόζουν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Η Επιτροπή Επασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και τη δική μας Επιτροπή Αναφορών εκπροσωπήσαν, εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, UNCRPD και η κυρία Φεραγκούτ και η κυρία Καβεσόν από κοινού εκπροσωπούν την Επιτροπή Αναφορών σε αυτή την ομάδα εργασία, σε αυτό το πλαίσιο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό που αυτή η Επιτροπή διόρισε δύο μέλη. Το περσινό έτος ήταν αρκετά έντονο σε σχέση με ζητήματα που σχετίζονται με αναπηρίες. Είχαμε την έκθεση Χέλγα Στίβενς που υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια με συνεισφορά από 10 επιτροπές και από τις ε, συνδεδεμένες επιτροπές ΠΕΤΗ και ΛΥΜΠΕ. Η δική μας επιτροπή έλαβε έναν μεγάλο αριθμό αναφορών από άτομα με αναπηρίες, τι οργανώσεις τους ή από άτομα που δρούν για το δικό του συμφέρον σε διάφορους τομείς. Φέτος το Σεπτέμβριο υλοποιήσαμε μια διερευνητική επίσκεψη στη Σλοβακία προκειμένου να διερευνήσουμε ισχυρισμού που έχουν να κάνουν με την κατάχρηση κονδυλίων από τα διορθωτικά ταμεία και επενδύσεις σε μικροπρόθεσμα ιδρύματα. Είχα την τιμή να προεδρεύω αυτή τη αντιπροσωπεία και συμποραίνω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το σχέδιο της έκθεσης με την λεπτομερή περιγραφή της επίσκεψης, καθώς και τα κύρια πορίσματα και οι κύριες συστάσεις θα παρουσιαστούν κατά τη σημερινή συνεδρίαση το απόγευμα. Είναι πολύ λογικό. Και Φυσικά, καθώς έχουμε τώρα αυτό το workshop, θα ακολουθήσουν τα πορίσματα της επισκεψής μας. Επίσης, εργαστήκαμε σκληρά στο φάκελο της συνθήκης του Μαρακές, κάτι που κρεμούσε για πολλά χρόνια. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που στις 30 Σεπτεμβρίου, μετά από μετά από τις 30 Σεπτεμβρίου, πάνω από 20 30 χώρες την έχουν επικυρώσει και πιστεύουμε ότι τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα και να κυρώσει τη συνθήκη του Μαρακές χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή. Στην Επιτροπή αυτή επίσης ε, γνωμοδοτούμε επί της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητα και η κυρία Κούνεβα, η οποία είναι ε, η συγγήτρια από την Επιτροπή Πέτη έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά και έχει ήδη καταθέσει 157 τροπολογίες, ενώ τα μέλη της Επιτροπής έδραξαν την ευκαιρία να βελτιώσουν περαιτέρω το κείμενο της Κομισιόν και εργάζονται επί περαιτέρω τροπολογιών. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα και θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Νομίζω ότι έχετε τώρα κάποια παραδείγματα για το τι κάνει η Επιτροπή μας σε αυτό το τομέα. πολιτικής. Και έχουμε ουσιαστικά σκεφτεί μια σειρά μέτρων για να παρουσιάσουμε, για να απαντήσουμε στις ε, αιτήσει που έχουμε. επίση θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη της Επιτροπής, αλλά του προσκεκλημένου μας, ε, να σκεφτούν επί του έργου που έχει γίνει καθόλου το έτος και τις δράσεις που πρέπει να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε και εμείς ως Επιτροπή αλλά και αυτό το θεσμικό όργανο. Με τη βοήθεια λοιπόν των εμπειρογνωμόνων και της κοινωνίας των πολιτών ελπίζουμε να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να απαντήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανησυχίες των πολιτών με αναπηρίες που πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τη Σύμβαση και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τώρα, θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο και αγαπητή φίλη Ρόζα Εστεράς Φεραγούτ, η οποία θα είναι συντονίστρια για το πρώτο πάνελ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πράγματι, περνάμε τώρα σε αυτό το workshop που αφορά πάρα πολλές ε, αναφορές που έχουμε λάβει από άτομα με αναπηρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους. Είναι εδώ και ο κύριος ε, Κώσα, ο οποίος ε, είναι πρόεδρος της Ομάδας για τις Αναπηρίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης έχει αναλάβει και να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της ομάδας προκειμένου τα άτομο με αναπηρία να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σεσίλια, η πρόεδρός μας, μας τα εξήγησε. Έχουμε ένα σημείο αναφορά που είναι η Σύμβαση του ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε και κατόπιν έχουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Αναπηρίες 2010-2020. Πέρσι τον Αυγουστό είχαμε μια συνεδρίαση στα Ηνωμένα Έθνη όπου έγιναν κάποιες παρατηρήσεις για το πώς είχε εφαρμοστεί η σύμβαση στα ευρωπαϊκά κράτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έγιναν λοιπόν κάποιες τελικές παρατηρήσεις, κάποιες συστάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή αυτής της σύμβασης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ πολλών παρατηρήσεων υπόθηκε ε, να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο παρακολούθησης της σύμβασης αυτής, συνέχεια της σύμβασης αυτής, δηλαδή ένα πλαίσιο για να ε, θέσουμε σε εφαρμογή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής Αναφορών Δηλαδή και εγώ και η κυρία να ε, συμμετέχουμε, συμμετέχει και ο συνήγορος του πολίτη. Συνήγορος είναι ε, ουσιαστικά πάρα πολύ, συμμετέχει πάρα πολύ, συμμετέχει και ο ΦΡΑ, Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, της αρχής, αν και κατόπιν ζητήθηκε να αποσυρθεί η Κομισιόν ε, προκειμένου να υπάρχει αντικειμενικότητα. Σε αυτό το πρώτο πάνελ, λοιπόν, θα παρουσιάσουμε τρεις μελέτες. Η πρώτη μελέτη θα παρουσιαστεί από τον Μάρκ Πρίστλεϊ, ο οποίος είναι καθηγητής και είναι υπερογνώμονας για θέματα με αναπηρίες. Θα μας κάνει μια παρουσίαση για το πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο εφαρμογής και με ποιο τρόπο η Επιτροπή Αναφορών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτουν σε εφαρμογή τη σύμβαση. Θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στο Μάρκ Πρίσλεϊ. Θα πω ότι είναι επιστημονικός διευθυντής ε, της ε, Ακαδημίας ε, των Εμπειρογνωμόνων για θέματα αναπηρίας. Επίσης είναι διευθυντής του Σχολείου Κοινωνικής και Πολιτικής Συνοχής, και Πολιτικής και θα μας παρουσιάσει αυτή τη μελέτη. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί όσοι είμαστε εντός του πλαισίου και εργαζόμαστε, ε, περιμένουμε να μας διαφωτίσει και ε, επίσης θέλουμε να εμβαθύνουμε και να βελτιώσουμε την εφαρμογή της σύμβασης αυτής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο και τη Συντονίστρια. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία της ε, ΠΕΤΗ γιατί ε, υποστηρίζει αυτή τη μελέτη και τη διαχειρίστηκε πολύ σωστά. Πιστεύω ότι πέρσι ε, αυτή την περίοδο παρουσιάσαμε το, την έκθεση η οποία ενημερώθηκε και μας δείχνει τις ε, εξελίξεις κατά το τελευταίο 12 καθώς και τις εξελίξεις, όπως είπε και η πρόεδρος ε, της δράσης του Κοινοβουλίου και την ανταπόκριση στη σύσταση των Ηνωμένων Εθνών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επιλέξω ορισμένα στοιχεία από την έκθεση. Η έκθεση αυτή δημοσιεύθηκε αρχικά το 2015 και μας δίνει ένα πλαίσιο και ανάλυση των δεδομένων με βάση τη Σύμβαση των ε, Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων και τον ρόλο της Επιτροπής. Υπάρχουν διάφορα κεφάλαια, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, για να κατανοήσουμε το ρόλο προστασίας και να δούμε και τις αναφορές που έλαβε ανά το χρόνο η Επιτροπή. Επιλέγουμε λοιπόν ορισμένες ε, αμφίσιμες ε, περιπτώσεις που έχουν προκαλέσει διαφορές σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τη δράση. Και προβάλλουμε και συστάσεις. Για να συνοψίσω Πέρσι μιλήσαμε για τα συμπεράσματα της έκθεσης και είδαμε ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αναπηρίας. Και επίσης υπήρξε μεγάλη υποστήριξη από το κοινό. Είχαμε ένα εκατομμύριο αναφορές, κάτι το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, κάτι το μοναδικό. Επίσης, αυτό το θέμα έθιξε ζητήματα διαχείρισης και διακυβέρνησης, καθώς και τον περιορισμό του ρόλου της Επιτροπής σας, διότι δεν μπορεί να προβάλλει δικαστική λύση. Και φυσικά έχουν γίνει και πολύ περισσότερα τον τελευταίο χρόνο. Και σας ευχαριστώ πολύ και για τις εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας που έχετε αναλάβει. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της μη δικαιοδοτικής ανταπόκρισης από τα κράτη-μέλη σε περίπτωση επίλυσης διαφορών. Και επίσης ορισμένα από τα δικαιώματα που θίγονται από τους πολίτες στις αναφορές δείχνουν τα όρια αρμοδιοτήτων νομικών αρμοδιοτήτων και πολλές φορές είναι δύσκολο να υπάρξει σωστή δικαιοδοσία από τα κράτη-μέλη. Επίσης, τα συμπεράσματα, τα περσινά συμπεράσματα έδειξαν ότι θα μπορούσαμε να προβάλλουμε ορισμένες διαδικασίες βελτιώσεων. Για παράδειγμα, θίξαμε το ζήτημα της υποβολής αναφορών στη νοηματική και επίσης πώς η γραμματεία, στα πλαίσια της γραμματείας, να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ε, σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και επίσης ομαδοποίηση αναφορών για να εστιάσουμε την προσοχή του κοινού σε θέματα αναπηριών. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μία ετήσια ανταπόκριση σε αυτές τις αναφορές και φυσικά η προστασία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτών των δικαιωμάτων. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 1 τέταρτο του εκλογικού σώματος έχει κάποια μορφή αναπηρίας, κάτι το οποίο δεν μπορούν να αγνοήσουν οι πολιτικοί. Είναι μεγαλύτερη σε ηλικία πολίτες και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτή η ε, κατηγορία. Πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν κύρια αξία της συνθήκης και η πρόεδρος μίλησε και για τη σημασία ύπαρξης μιας διεθνούς συνθήκης σε σχέση δηλαδή με την κάλυψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε καλύψει μέχρι τώρα και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα διευθετηθεί. Έτσι ώστε να ε, προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς και παγκοσμίως και εμείς να αποτελέσουμε την εμπροστοφυλακή. Άρα, στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχει ένα εγχώριο πλαίσιο εφαρμογής ε, αυτών των δεδομένων σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Και από όσο γνωρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα εγχώριο πλαίσιο. Αλλά φυσικά δεν υπάρχουν τα ίδια θεσμικά όργανα και οι ίδιες αρμοδιότητες. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ένα ε, ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δούμε λοιπόν τις αλλαγές που έχουν επέλθει, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με πέντε σώματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηριών. Και τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν ότι ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσυρθεί από αυτό το πλαίσιο όσον αφορά θέματα ανεξάρτητης ερμηνείας και γι' αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη ερμηνεία του άρθρου 33 από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών όπου ακριβώς αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι μηχανισμοί προστασίας και εποπτείας. Υπήρξαν διχογνωμίες κατά πώς αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητοι μηχανισμοί ή αυτόνομοι μηχανισμοί ή όχι. Το θέμα είναι σχετικά περίπλοκο, αλλά η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία έχει αποσυρθεί από το επίσημο αυτό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, αν και δεν έχει γίνει και ε, τυπικά γραπτός. Αυτό τι σημαίνει ως προς την προστασία. Όπως είπαμε και πέρσι, τότε υπήρχαν διάφοροι μηχανισμοί προστασίας μέσα στα πλαίσια αυτής της πλαισίωσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει η διαδικασία αναφορών όπου οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να υποβάλει αναφορά. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει αυτό το ρόλο ως προς διοικητικά θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης Επίσης, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηριών λαμβάνει πολλές αιτήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία επίσημη δομή προσφυγών και καταγγελιών που δεν εντάσσεται απόλυτα σε αυτή την ε, πλαισίωση. Γι' αυτό έχει σημασία να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συντονισμός αυτών των φορέων για να υπάρξει ένας ενιαίος μηχανισμός προστασίας. Όπως είπα, ε, υπήρξαν αλλαγές ως προς την ε, συμμετοχή και τη διαχείριση. Έχουμε μία ιστοσελίδα εργασίας στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και αυτό φαίνεται και από την επίσημη ιστοσελίδα. Η πρώτη σελίδα δεν έχει ενημερωθεί σε σχέση με τη δεύτερη και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα εργασίας το οποίο επικαιροποιείται και είχαμε και σχόλια από διάφορους φορείς για το ρόλο και την εξέλιξη του δικτύου και προσπαθήσαμε να διευρύνουμε και το πλαίσιο προστασίας μετά από συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Και η ΦΡΑ ζήτησε μία γνωμοδότηση για νομική βάση για να μπορέσουμε να δράσουμε σωστά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν Υπάρχουν ενδιάμεσες διευθετήσεις και οργανώσεις. Η ΦΡΑ προβάλλει και τη, τη γραμματιακή υποστήριξη όπου σε μία ιδεώδη κατάσταση πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Έχουμε λοιπόν, βρισκόμαστε σε μία ενδιάμεση φάση η εξέλιξη. Ζητώ συγγνώμη γιατί χρειάστηκε να παραλείψω ορισμένες διαφάνειες. Επίσης, όπως είπε και η Πρόεδρος, μιλάμε και για το ρόλο της Επιτροπής σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Τώρα, ως προς τις ίδιες ε, τις ε, αναφορές. Ο ρόλος προστασίας της ΠΕΤΗ είναι πολύ σημαντικός γιατί λαμβάνει αναφορές εδώ και αρκετά χρόνια και σχετικά με αναπηρίες που είναι ένα βασικό θέμα. Κάτι το οποίο παρακολουθούμε. Σε σχέση με το γράφημα που είδαμε πέρσι βλέπουμε και κάτι παράλληλο, δηλαδή ως προς την προσβασιμότητα και την κοινωνική προστασία, εδώ έχουμε να κάνουμε με τα δύο βασικότερα θέματα. Ως προς την προσβασιμότητα έχουμε μια αύξηση αναφορών, ενώ πέρσι το, πιο, το βασικότερο θέμα ήταν η κοινωνική προστασία. Μας ενδιαφέρει και η ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας, η οποία τώρα συζητείται, και βλέπουμε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Άρα έχουμε την προσβασιμότητα καταρχήν, την ανεξαρτησία κατά τη διαβίωση, τα δικαιώματα κατά την εργασία και την κοινωνική προστασία. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει και μία σαφής νομική βάση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε αυτά τα παραδείγματα πέρσι και θα ήθελα να μιλήσω για τα πλέον πρόσφατα ως προς το θέμα της νοηματικής που είναι ένα από τα βασικά θέματα γιατί είχαμε μία αίτηση από την Ένωση Κοφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε ότι οι αναφορές που θα έχουν επιτυχία είναι αυτές που έχουν συνταχθεί σωστά και την χάνουν συλλογικής υποστήριξης κοινωνικά. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία αναφορά που στάθηκε και στην περσινή σύσταση, δηλαδή μία πολύ απλή αναφορά και η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αναφορές και στη νοηματική το εξετάσαμε αυτό το επιμέρους ζήτημα, θεωρήσαμε ότι αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι να υπάρχει και μία άλλη λειτουργία στην ε, πύλη, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει και ψηφιακή μορφή υποβολής της αναφοράς και φαίνεται ότι αυτή η πύλη είναι έτοιμη. Βλέπετε λοιπόν εδώ την πύλη και την ιστοσελίδα που λέει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διάφορες μορφές, δηλαδή ε, MP3, MP4, PNG, ε, DOCS και ούτω καθεξής και MPEG. Και ε, αυτό σημαίνει ότι οι αναφορές πρέπει να υποβληθούν και μπορούν να υποβληθούν και σε αυτή τη μορφή. Το θέμα είναι ένα θέμα συζήτησης. Ένα τελικό ζήτημα που θα ήθελα να θίξω αφορά τη, τους περιορισμούς της πλαισίωσης. Οι διάφοροι φορείς μιλήσαν για τους περιορισμούς της εντολής αυτής. Δηλαδή το κάθε μέσον και φορέας λειτουργεί με τη δική του εντολή. Όπως ε, είπε και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΦΡΑ, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας και να μπορεί να υποβληθεί μία αναφορά μέσα στα πλαίσια μιας ενιαίας μορφής ε, παρουσίασης. Επίσης δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε ένδικα μέσα, όπως μας τόνισε και το Φόρουμ Αναπηριών. Και θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια των αρχών των Παρισίων. Εδώ δεν σας προβάλλω συστάσεις, είναι θέματα προσυζήτηση. Οι αρχές των Παρισίων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρονται στα εθνικά κοινοβούλια τα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για μια πλουραλιστική προσέγγιση όπου να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των κοινοβουλίων στις αρχές αυτές και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό. Και πολλά κράτη δεν έχουν Ινστιτούτα Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που να ακολουθούν αυτό το μοντέλο προστασίας των αναπηριών. Δεν υπάρχει δηλαδή ε, πλουραλιστική προσέγγιση με συμβουλευτικές αρχές και συνεισφορά του ακαδημαϊκού κόσμου. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί τρόποι για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ίσως ε, θα ε, υπάρξει μεγαλύτερος γραφειοκρατικός φόρτος κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα με αυτό το θέμα το οποίο έχει οδηγήσει και σε διχογνωμίες. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι αυτό που μας είπατε είναι ενδεικτικό. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το πλαίσιο για να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες του πλαισίου περνάμε στην επόμενη... Τον επόμενο ομιλητή, Σέσσαρα Μύρες Μόντες, ε, είχε συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και αφορά τη σύμβαση του Μαρακές, η οποία εγκρίθηκε από μάλλον στο Μαρακές εδώ και τρία χρόνια, το 2013, έτσι ώστε να υπάρχουν ε, διασυνοριακές ανταλλαγές οπτικοακουστικών μέσων, βιβλίων και ούτω καθεξής μέσα στα πλαίσια της ε, τήρησης των πνευματικών δικαιωμάτων έτσι ώστε οι άνθρωποι με αναπηρίες να έχουν αυτή την προσβασιμότητα. Και να ε, καταξιωθεί. Όπως ξέρετε, τον Απρίλιο του 2014 η Ένωση κύρωσε αυτή τη σύμβαση, αλλά επειδή υπάρχουν θέματα αρμοδιοτήτων, το θέμα έχει κάπως παγώσει και τέλος, το Μάιο του 2015 το Συμβούλιο υπέβαλε έτοιμα προς την Επιτροπή για να συντάξει μία οδηγία για να τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση του Μαρακές. Και η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση οδηγίας εδώ και μερικούς μήνες και στόχος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, ε, μουσικών ε, παρτιτούρων και ούτω καθεξής. Και θα δούμε και σήμερα το απόγευμα στις αναφορές μας ότι πολλές αναφορές αναφέρονται στη συνθήκη του Μαρακές. ο δόκτωρ Σέσαρα Ραμίρες Μόντες, ο οποίος είναι συντονισμός του Εράσμους στη ε, νομική σχολή, θα μας μιλήσει για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ψηφιακής μορφής για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε και αυτή την οδηγία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να διευκρινίσω το εξή. Είμαι στο Πανεπιστήμιο του Λίτσα, αλλά σπουδάζω στην Οξφόρδη. Αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσω. 15 λεπτά έχω μόνο στη διάθεσή μου και το αντιλαμβάνομαι για να παρουσιάσω την ε, <clears throat> έκθεσή μας, την ε, έρευνά μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω εντάχει τα βασικά σημεία. Για να σας δώσω μια ιδέα για τη μεθοδολογία που ακολουθούμε. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια εμπειρική έκθεση, μελέτη. Προετοιμάσαμε λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο και μοιράσαμε στα μέρη του Συμβουλίου. Θέλουμε να διαπιστώσουμε τους ε, λόγους που οδήγησαν το μπλοκάρισμα της επικύρωσης ε, της συνθήκης της Μαρακές. Ε, δέκα ερωτήσεις λοιπόν στείλαμε και να σας πούμε ότι λάβαμε μία απάντηση και ουσιαστικά δεν απαντηθήκε καμία ερώτηση. Κοιτάξαμε λοιπόν τις πρωτογενείς πηγές, την νομολογία και τις ακαδημαϊκές τοποθετήσει, μεταξύ άλλων και τα έγγραφα πολιτικής. Αυτά λοιπόν τα κάναμε για να συντάξουμε την έρευνα αυτή. Και αυτό είναι το περιεχόμενο λοιπόν της ε, έρευνας, της έκθεσης ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει το πλαίσιο, αν θέλετε, της συνθήκης του Μαρακές. Εδώ διαπιστώνουμε ένα κοινωνικό κίνημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ε, πλατφόρμα για αυτή την ε, ιστορική σύμβαση. Στη συνέχεια περνάμε στην περιγραφή των θεμελιωδών ανθρωπινών δικαιωμάτων που είναι η πρόσβαση στον πολιτισμό και στην πληροφορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ήταν θεμελιώδες στις προτάσεις που κατατέθηκαν από την Οργάνωση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Από το 2003 και μετά η Ένωση Τυφλών προσπάθησε να προωθήσει μια τέτοια πρόταση σύμβαση που τελικά κατέληξε στη συγκεκριμένη πρόταση του 2009 από την οποία και αναδείχθηκε η συνθήκη του Μαρακές. Η συνθήκη του Μαρακές στη συνέχεια εξηγούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει οι τέσσερις βασικές προδιαγραφές στο σημείο 4 της ε, έκθεσης και επίσης τονίζουμε στην έκθεση αυτή καταρχάς τη μοναδική φύση της συνθήκης αυτής και κατά δεύτερον το γεγονό ότι είναι η πρώτη διεθνή συνθήκη που συνδυάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα των αναπηρών και τα δικαιώματα πνευματική συντεκτησίας, ιστορική σημασία. Τέτοια διεθνή σύμβαση. Στη συνέχεια, προβαίνουμε σε κάποια καταληκτικά σχόλια που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την επικύρωση σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Και αυτό είναι βασικό θέμα σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της, του Μαρακές. Γιατί? Γιατί ένα από τα βασικά επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαν τα κράτη-μέλη για το γεγονός ότι δεν επικυρώνουν την συνθήκη του Μαρακές ήταν ότι η, συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να τροποποιήσει τα δικαιώματα Πνευματική ιδιοκτησία και τη σχετική νομοθεσία. Και το θέμα ήταν επίσης, ε, το επιχείρημα μάλλον που χρησιμοποιήθηκε ήταν επίση και το θέμα τη ε, μεικτή αρμοδιότητα και των αντικρουόμενων ε, αρμοδιοτήτων. Και τέλος, συστάσει προ το Κοινοβούλιο, προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προ τα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν περιλαμβάνει συνοπτικά η έκθεση, η μελέτη. Τώρα, θα ήθελα εντάχει να σας εξηγήσω ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο. Η ανάγκη για ένα διεθνές πλαίσιο, μια διεθνή συμφωνία που θα προβλέπει υποχρεωτικές εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών και των ατόμων που δεν μπορούν να αναγνώσουν δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή από τη δικασία του 80. Άρα η συνθήκη του Μαρακές δεν αναφέρεται σε κάποια καινούργια ανάγκη. Οι ανάγκε αυτές ε, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στη μελέτη μας λοιπόν ε, καταγράφουμε την ιστορική αυτή διαδρομή και τα αίτια που οδήγησαν στην ε, σύμβαση αυτή. Κάτι άλλο που περιλαμβάνεται στο τμήμα αυτό. Όπως είπε σωστά και η Πρόεδρος, εντοπίζεται το θέμα της Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που εγκρίθηκε το 2006. Ορόσημο. Ορόσημο αποτέλεσε αυτή η σύμβαση και σημαντική όθηση για την πρόταση για τη συνθήκη του Μαρακές. Γιατί πέρα από το ότι εγγυάται βασικά θεμελιώδη ανθρωπίνα δικαιώματα για τους αναπηρούς βάσει του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία όπου δηλώνεται ότι η αναπηρία περιλαμβάνει κοινωνικά ουσιαστικά εμπόδια. Για πρώτη φορά υπάρχει αναγνώριση του γεγονότος ότι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων ενδεχομένω να οδηγεί σε φραγμούς, σε εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία. Άρα δημιουργείται υποχρέωση για τις χώρες που προσυπογράφουν να καταργήσουν τα εμπόδια αυτά. Άρα παρακολουθούμε τις ιστορικές ε, ρίζες και τα αίτια Τη σύμβαση και είναι βασικό εδώ. Είναι βασικός ο ρόλος των υπηρεσιών του ΟΗΕ, προκειμένου αφενός να υπάρχει καλύτερη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πολυμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες, όπου και διευκρινίζεται η Συμφωνία TRIPS, για παράδειγμα, το 1994 και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των πνευματικών δικαιωμάτων, τη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου για την προστασία των διεθνών των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, από πλευρά των αναπτυγμένων χωρών, που τελικά οι αναπτυσσόμενες χώρες δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερως να συμμορφωθούν με αυτές τις υποχρεώσεις τους. Και να διευκρινίσουμε ότι η πλειονότητα των ατόμων που είναι τυφλά και δεν μπορούν να διαβάσουν είναι από τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Μόνο το 1 τέταρτο των βιβλίων και των εντύπων μπορούν να διδεθούν στα άτομα αυτά στις αναπτυσσόμενες χώρες. 1% μόνο, συγγνώμη, ε, έχουν στην διάθεσή τους. Και άρα ο ρόλος του ΟΗΕ είναι να τονίσουν ακριβώς το χάσμα αυτό που υπάρχει μεταξύ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και των θεμελιωτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί στη συνέχεια τα δικαιώματα των αναπήρων εντοπίστηκαν ως βασικό θέμα σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και έτσι δόθηκε ένα πλαίσιο για πρώτη φορά όπου συναντιούνται πολύ διαφορετικοί τομείς του δικαίου, της νομοθεσίας και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των αναπήρων. Και περνάμε γρήγορα γρήγορα σε κάποια ανάλυση που έγινε από τις υπηρεσίε του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πρόσβαση στον πολιτισμό, στην επιστήμη. Στο άρθρο 15 της σύμβασης περιλαμβάνονται όλα αυτά. Στο σημείο λοιπόν αυτό, τι διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε πώς γίνονται παραλληλισμοί από τον ΟΗΕ για το δικαίωμα πρόσβαση στον πολιτισμό και την υποχρέωση του άρθρου 15 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για να καταργηθούν οποιοδήποτε φραγμή και εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Άρθρο 21 και άρθρο 30. Συνδυαστικά της σύμβασης. Εδώ λοιπόν δίνουμε κάποια παραδείγματα για το τι λένε οι υπηρεσίε αυτές. Τονίζουν ότι η πρόσβαση στην, ε, στον πολιτισμό και στα πολιτισμικά αγαθά προϋποθέτει και την διάσταση της ε, προσβασιμότητας. Ότι δεν υπάρχει νόημα να υπάρχουν τα δικαιώματα αυτά εάν δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά και τα άτομα με αναπηρία. Εντόπισαν λοιπόν και την διάσταση της ε, προσβασιμότητας, την οποία και τονίζουμε και εμείς στην έκθεση. Εκ παραλληλού, επειδή υπάρχει αυτή η αντίφαση μεταξύ των ε, πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ε, τονίζουμε και την μηνιαμελαστική προσέγγιση. Τελικά, αυτή η διατύπωση, αυτές οι συνθήκες είναι που έδωσαν την τελική όθηση, προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα πνευματικά δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν ε, ε, ακτιβιστές για το θέμα της επιστήμας σε διεθνές επίπεδο. Και οι ακτιβιστές αυτοί προωθούν λοιπόν τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην ε, και έχουμε και την ατζέντα αναπηρίας. Όλα αυτά λοιπόν συγκλίνουν προκειμένου να διαμορφώσουν το πλαίσιο το οποίο τελικά οδήγησε στις προτάσεις αυτές και αναλύσαμε τις προτάσεις στο σημείο αυτό. Τέσσερις προτάσεις λοιπόν έγιναν αρχικά. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μία από τις πιο παροχημένες Λύσεις για τα δικαιώματα των αναπήρων είναι η πρόταση τη ευρωπαϊκή ένωση και τον είπα παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά είχαν σχετική υποχρέωση υπό τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε μια σύσταση, οι ΙΠΑ ζήτησαν απλά ένα κοινό εργαλείο, μια κοινή συμφωνία. Η Παγκόσμια Οργάνωση Τυφλών έκανε μια πρόταση με μια ομάδα χωρών Λατινικής Αμερικής και ζήτησε την ε, υποχρεωτική, τον υποχρεωτικό περιορισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να υπάρχει τέτοια προσβασιμότητα. Ζητήθηκε λοιπόν να είναι δεσμευτικές, υποχρεωτικές αυτές οι δεσμεύσεις, αυτές οι εξαιρέσεις. Να υπάρχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο, μια διεθνώς ε, δεσμευτική σύμβαση. Εμείς εξηγούμε λοιπόν τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Και ένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης αυτής είναι το εξή. Εντοπίστηκε ένα ευρύ πλαίσιο των δικαιούχων και τονίστηκε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει εμπορική διαθεσιμότητα ως προϋπόθεση η Διεθνή Ένωση Τυφλών και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών εντόπισαν σε σχετικές έρευνες της Επιτροπής ΠΕΤΗ το 2009 ότι ως τότε ουσιαστικά αγνοούνταν παντελώ οι ανάγκε των τυφλών. Τόνιστηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για εμπορική διαθεσιμότητα γιατί δεν θεωρούνταν εμπορικός ε, κερδοσκοπικές Περνάμε λοιπόν στη συνέχεια στη συνθήκη του Μαρακές. Η συνθήκη του Μαρακές λοιπόν. Ο σκοπό έχει την εισαγωγή των υποχρεωτικών αυτών εξαιρέσεων στο δίκαιο, στην νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα από πλευρά των κρατών μελών, προκειμένου να επιτρέπεται η διασυνοριακή ανταλλαγή τέτοιων αντιτύπων. Σε αντίθεση με άλλες συμβάσεις, του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικών Δικαιωμάτων. Για πρώτη φορά εδώ δημιουργείται το δικαίωμα, το υποχρεωτικό δικαίωμα χρήσης. Όχι τόσο δικαιώματα δηλαδή των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων, όσο των χρηστών. Και υπάρχει έτσι η δυνατότητα διασυνοριακής ανταλλαγής των δικαιωμάτων αυτών και των αντιτύπων αυτών. Βλέπουμε λοιπόν τι προβλέπει η συνθήκη τη Μαρακέ. Τέσσερις βασικές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι στο άρθρο 4.7 υποχρεωτική ε, φύση των εξαιρέσεων αυτών. Εξαιρέσει για το δικαίωμα αναπαραγωγή, διαθεσιμότητα, διανομής. Πρόκειται για αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνονται στο copyright και τα βλέπετε στο κείμενο, αλλά προβλέπετε και υποχρέωση για τα κράτη-μέλη για να αφαιρεθούν οποιαδήποτε τεχνολογικά μέτρα προστασίας. Αυτό ήταν ε, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε για πολύ καιρό τα πολλούς ανθρώπους. Κρυπτογράφηση, συστήματα κλειδώματος τέτοιων ε, περιεχομένων. Περιλαμβάνουμε λοιπόν ποιες είναι οι βασικές υποχρέωσεις και στη συνέχεια περνάμε Μάλλον πριν περάσω στο επόμενο σημείο, να πω το εξή. Στο σημείο αυτό εξηγούμε γιατί προέκυψε αυτή η διαφωνία σε ό,τι αφορά την επικύρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. όπω είπε η πρόεδρο, 30 Σεπτεμβρίου του 2016 τέθηκε σε εφαρμογή η συνθήκη. Και ο Καναδά έγινε η 26η χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη. Πάνω από 100 χώρες έχουν υπογράψει, αλλά μόνο 26 έχουν προσυπογράψει ως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικυρώσει, δεν έχει επικυρώσει ακόμα την ε, σύμβαση. Και το θέμα λοιπόν είναι ε, το θέμα της ε, χρονικής συγκυρίας. Πότε θα γίνει η επικύρωση. Και το θέμα είναι και η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το copyright. Εμεί τονίζουμε ότι μπορεί να γίνει επικύρωση χωρί να υπάρχει αυτόματη υποχρέωση προ... προσαρμογή του συστήματο copyright. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε λοιπόν να απευθύνει ερώτημα προ το δικαστήριο για να ζητήσει τα θέματα αρμοδιότητας. Ο Γενικός Εισαγγελέας δημοσίευσε την άποψή του στι 8 Σεπτεμβρίου του τρέχοντο έτου, αν και δεν έχει αποφανθεί ακόμα το δικαστήριο. Ο Γενικό Εισαγγελέα ήταν ευνοϊκό σε ό,τι αφορά την νομική αρμοδιότητα της Ένωσης και έθεσε το θέμα της νομικής βάσης. Και αποφάνθηκε ότι η συνθήκη του Μαρακές θα αλλάξει σημαντικά ένα τμήμα του κοινωτικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θεωρεί ότι θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και θα μπορούσε να ακολουθήσει το άρθρο 3 της ε, συνθήκης. Εδώ λοιπόν κάνουμε κάποιες συστάσεις προς το Κοινοβούλιο και ζητούμε από το Κοινοβούλιο Ιδιαίτερος να ασκήσει πίεση για την ταχεία επικυρώση. Ζητούμε από το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας και τη Σχετική Συμμαχία Αναπήρων σε ό,τι αφορά και άλλα υπόθετα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συστήνουμε να συνεχίσει η διαδικασία επικύρωση και να σκεφτεί πίεση προ την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και την πολύ ευνοϊκή γνωμοδότηση του Γενικού Συγγελέα. Δεν είναι δεσμευτικό αυτό ασφαλώς, αλλά κατά 95% ακολουθείται από το δικαστήριο η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα και αυτό είναι υπέρ τη αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε και κάποιε συστάσει προ τα κράτη-μέλη. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν και να συνεργαστούν επικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτή. Δύο προτάσει: Μία για μία οδηγία και μία για ένα κανονισμό. Και το καλό είναι ότι οι προτάσει αυτέ ε, προβλέπουν τι βασικέ διδάξεις τη συνθήκη του Μαρακέ. και χρησιμοποιούν τις ρήτρες exception plus, δηλαδή εξαιρέσεις συν. Μπορεί να πάμε και πιο πέρα από το Μαρακές, δηλαδή το Μαρακές προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο, αλλά επιτρέπει στα κρατημέλη να πάνε και παραπέρα. Προτείνεται λοιπόν ένα περιορισμό και άλλων δικαιωμάτων. Μπορούμε να πάμε και πιο πέρα όμω. Ενθαρρύνουμε τα κρατη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσου εργάζονται με ομάδε ε, ατόμων με αναπηρία να βρουν ποιε είναι οι ανάγκε, ποια άλλα ανθρώπινα δικαιώματα περιορίζονται και θα πρέπει να βελτιωθούν. Κάνουμε λοιπόν μια σειρά συστάσεων στο σημείο αυτό. Και κάτι που λείπει στο σημείο αυτό είναι το εξή. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει το πώς μπορούν να επιτευχθούν στην πράξη οι στόχοι της συνθήκης του Μαρακές. Να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, α, α, αγωγών και συλλογικών αγωγών από πλευρά τη συνθήκη του Μαρακέ, να υπάρχει ένα σχέδιο δράση για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, για να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχο προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του Μαρακές, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη, ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ. Pues muchas, muchas gracias. Σας ευχαριστούμε. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της ομάδας ε, για τις ανεπηρίες ε, θα διαβιβάσουμε αυτή την αναγκαιότητα να πιέσουμε για να υπάρξει έγκαιρη κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε στην τελευταία ομιλήτρια αυτού του πρώτου πάνελ, η κυρία Καμίλα Πάρκερ, και θα μας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με ποιο τρόπο τα ευρωπαϊκά διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία μπορούν να υποστηρίξουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να μπορούμε να φτάσουμε στην ένταξη. Στην περίοδο 2007-2013 πολλές φορές ε, τα ταμεία δεν παρουσίασαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι η νέα ρύθμιση για τα ταμεία το 2013-2020 ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε οποιοδήποτε κόστος, αλλά μόνο με την εγγύηση του θα υπάρξουν αποτελέσματα και ότι αυτά πρέπει να συνάδουν με τη στρατηγική 2020, εκπαίδευση, καινοτομία, βιωσιμότητα και φυσικά και μη αποκλεισμού, έτσι ώστε να έχουμε αηφόρο και φυγή ανάπτυξη. Θα μας μιλήσει λοιπόν ε, μιλήτρια για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ταμεία για να μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα της ένταξης ε, και όχι μόνο στην καθημερινότητα αλλά και στην εκπαίδευση. Δηλαδή η εκπαίδευση είναι συμμετοχική. Επίσης και στην απασχόληση αλλά και στη ζωή, στην κοινότητα. Και αυτό το ανέφερε και η Σύμβαση, να μπορούν να ζουν τα άτομα σε κοινότητα και να δούμε την διαφορετικότητα ως κάτι θετικό που μας εμπλουτίζει όλους. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Καμίλα Πάρκερ για να μας μιλήσει για αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Είναι ουσιαστικά μία από τις ε, ιδρύτριες ε, ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Μετσοτή Ζωή και είναι ουσιαστικά και δικηγόρος που υπερισπίζεται τα άτομα με αναπηρίες. Παρακαλώ Καμίλα. Σας ευχαριστώ. θα κάνω μια παρουσίαση εγώ αλλά και συνάδελφος, η Νέα Συμβουλή. Εγώ θα ξεκινήσω. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την έκθεσή μας. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το πλαίσιο. Εξετάζουμε την κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία και τις συγκεκριμένε ανησυχίες ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους με αναπηρία που ζουν μέσα σε ιδρύματα εδώ σε όλη την Ευρώπη και εξετάζουμε το σημαντικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Διευθυντικών και Επενδυτικών Ταμείων στο να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αυτά τα ταμεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για να βοηθήσουν ένα κράτος μέλος να πετύχει τη μετάβαση από ε, την μέρημνα σε ιδρύματα στην ζωή, στην κοινότητα. Να υποστηρίξει δηλαδή την υποστήριξη εναλλακτικών τη δημιουργία εναλλακτικών και να παράσχει και τεχνική υποστήριξη στα κράτη-μέλη για να πετύχουν μια πολύπλοκη διαδικασία σε ό,τι αφορά την αποϊδρυματοποίηση. Είχαμε μια σειρά εκθέσεων που τόνισαν την τεράστια ανησυχία για τη χρήση των διαθροτικών ταμείων στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την επένδυση σε ε, μέρημνα σε ιδρύματα και αν και τονίστηκε η σημασία της ε, κοινωνικής συμπερίληψης, ε, υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να συνεχιστούν κάποια προβλήματα. Ένα μέρος της εκθεσής μας ε, τόνιζε τα δυνάμει προβλήματα για τα μελλοντικά έτη χρήση των διαφορετικών ταμείων και είναι γιατί είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται για να διατηρηθεί αυτή η μέρημνα στα Ιδρύματα. Θα σας ε, εξηγήσω τι σημαίνει ο όρος community living, ε, ζωή στην κοινότητα. Χρησιμοποιείται ο όρος αυτός για να διασφαλίσουμε όταν μιλάμε για τη ζωή στην κοινότητα και τη μετάβαση από την ιδρυματική μερίμνα στη ζωή στην κοινότητα. Εξηγούμε ότι δεν πρόκειται απλώ ε, για θέμα μεταφοράς των ανθρώπων σε περιβάλλοντα που είναι βελτιωμένα. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν υποστήριξη και υπηρεσίες οι άνθρωποι που τους βοηθούν να συμμετέχουν σε αυτή την κοινότητα, να πάνε στη δουλειά τους, ε, στην εκπαίδευση και να τονίζουν τη σημασία της κοινωνικής ε, συμπερίληψης. Αυτό τονίζεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 19 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Εκεί αναφέρεται το δικαίωμα να ζει κάποιος ανεξάρτητα και να συμμετέχει στην κοινότητα. Ο στόχος της μελέτης ήταν να τονίσει την πιθανή χρήση των Ευρωπαϊκών Διευθυντικών και Επενδυτικών Ταμείων στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να ζουν στην κοινότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους σε ιδρύματα. Έτσι λοιπόν, ε, τονίζουμε τα βήματα που μπορούν να γίνουν για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα διευθυντικά ταμεία προς αυτό το σκοπό και να διασφαλίσουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται για να συντηρήσουν, να διατηρήσουν την ιδρυματική μέρημνα. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για κάποιες ε, αιτίες που προκαλούν ανησυχία. Συνεχίζει να υπάρχει υψηλό αριθμός ατόμων με αναπηρίες σε όλη την Ευρώπη σε ιδρύματα. Πολλές εκθέσεις ε, κατήγγυλαν τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα ιδρύματα αυτά. Υπάρχει ένα σύστημα επιτροπία σε πολλές από αυτές τις χώρες. Ουσιαστικά αφαιρεί το δικαίωμα των ανθρώπων να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και αυτό είναι μια πολύ δύσκολη και σημαντική πτυχή της τοποθέτησης σε ίδρυμα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ε, ουσιαστικά δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις και άλλοι αποφασίζουν για το που θα ζουν και αν θα συνεχίσουν να παραμένουν σε ιδρύματα. Έτσι λοιπόν, αυτός ο συνδυασμός της ιδρυματοποίησης και της επιτροπίας αντίκειται στο στόχο ότι όλα τα κράτη-μέλη που έχουν θέσει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι να μπορούν να ζουν όλοι οι άνθρωποι στην κοινότητα. Και άλλη μια μεγάλη ανησυχία είναι ότι υπάρχει ανεπαρκής προσοχή στο ζήτημα αυτό. Αν δούμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν λίγες πληροφορίες για ανθρώπους με αναπηρίες. Επίσης, δεν έχουν αναπτυχθεί υπαρκώ οι υπηρεσίες που βασίζονται στη ζωή στην κοινότητα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, για να μπορούν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν εναλλακτικέ. Όμως, εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι αν και τα κράτη-μέλη έχουν δηλώσει ότι θέλουν να προχωρήσουν προς αυτή τη μετάβαση, είναι πολύ αργή η διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που τονίζεται από την Επιτροπή στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Εξετάστηκαν μία σειρά κρατών και εξετάστηκε πώς ε, υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους τα κρατή μέλη στα πλαίσια της Σύμβασης η Επιτροπή μελέτησε μία σειρά εκθέσεων που αφορούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε ότι η Επιτροπή τόνισε κάποιες σημαντικές ανησυχίες σε τρεις τομείς. Καταρχήν, ότι οι αριθμοί των ατόμων που ζουν σε ιδρύματα θα να, έχει, να έχουν αυξηθεί. Αυτό είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορά μόνο τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά Βρίσκουμε αυτή την κατάσταση και σε άλλα κράτη, δηλαδή ότι τοποθετούνται περισσότεροι άνθρωποι σε ιδρύματα. Η Επιτροπή επίσης τόνισε το γεγονός ότι συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη ε, υπηρεσιών που βασίζονται στη ζωή στην κοινότητα και επίσης τόνισε το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία Τη μετάβαση ε, από την ιδρυματική μέρημνα στη ζωή στην κοινότητα. Έτσι λοιπόν η διαδικασία της αποϊδρυματοποίηση που λένε τα κράτη-μέλη ότι έχουν θέσει σε εφαρμογή, σε πολλές περιπτώσεις δεν προχωρά σε επαρκές επίπεδο. σε σχέση με τη χρήση τώρα των διορθωτικών ταμείων, γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό. Γιατί Αυτά τα ταμεία δίνουν στη δυνατότητα στα κρατημέλη να κάνουν αυτή τη σημαντική μετάβαση από τα παλιά συστήματα στο να αναπτύξουν εναλλακτικέ υπηρεσίες που προωθούν τη ζωή στην κοινότητα και την συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Τι είδαμε στο παρελθόν πολύ συχνά. Τα ευρωπαϊκά διαφορετικά ταμεία έχουν χρησιμοποιηθεί για να γίνουν επενδύσεις σε ιδρυματική μέρημνα. Ενίοτε χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για την ανακαίνιση των ιδρυμάτων, αλλά και για να υπάρξει και επέκταση των κτηρίων. Είναι δύσκολο να βρούμε πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί σε αυτό το τομέα και οι πληροφορίες, κυρίως από την κοινή των πολιτών, υποδηλώνουν ότι στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Λετωνία, στη Λιθουανία και στη Ρουμανία και Τη Σλοβακία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε ιδρυματική μέρημνα. Αυτό δεν ε, σημαίνει μόνο ότι διατηρείται η ιδρυματική μέρημνα, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να έχουν, ε, μην έχουν χρησιμοποιηθεί χρήματα για την ε, ανάπτυξη εναλλακτικών. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ενώ κάποιες υπηρεσίες φαίνεται να προωθούν τη ζωή στην κοινότητα, στην πραγματικότητα τι κάνουν. Υποστηρίζουν υπηρεσίες που συνεχίζουν τον πολιτισμό της ιδρυματικοποίησης, δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά καθεστώτα και συνεχίζουν να αποκλίνουν ανθρώπους που ζουν στις εγκαταστάσεις αυτές από το να έρθουν σε επαφή με τον εξωκόσμο και από το να έχουν ευκαιρία να συμμετέχουν στην τοπική ζωή της κοινότητας υπάρχει ένας ε, όρος, ε, όπως αναφέρεται σε μίνι ιδρύματα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδυλία για κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι πάλι κάτι που τονίστηκε από την Επιτροπή τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατομών με, με αναπηρία σε αρκετέ χώρε. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να επενδύουν σε ιδρυματική μέρημνα. Και πάλι, δεν πρόκειται απλά για χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Συμβαίνει σε μια σειρά χωρών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους τομείς που ανησυχούν ιδιαίτερα την Επιτροπή είναι το θέμα ότι χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να διατηρηθεί η ιδρυματική μέρημνα και αναφέρθηκε η Επιτροπή σε μια σειρά χωρών και το τόνισε ω ένα θέμα μεγάλης ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το επιλύσει αυτό το θέμα και να προωθήσει την αποϊδρυματοποίηση. Αν δούμε λοιπόν τη σημερινή προγραμματική περίοδο, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε το εξής. Το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί ότι δεν θα πρέπει πλέον τα ευρωπαϊκά κονδύλια να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ιδρυματικής έρευνας, αλλά αν δείτε την πρόοδο σε μία έκθεση που αναφέρεται πώς σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα κρατημέλη, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο ξεκολουθεί να υπάρχει έλλειψη οράματο ε, για τη ζωή στην κοινότητα. Αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν θέτουν ένα σαφέ όραμα για τη ζωή στην κοινότητα για του ανθρώπου με αναπηρίε. Και πολύ συχνά αφήνουν κάποια άτομα εκτό, κάποιε ομάδε ατόμων εκτό. Και επίση, αν δούμε και το σχέδιο δραστηριοτήτων, φαίνεται ότι συνέχιζε να υπάρχει σχεδιασμό για επένδυση σε ιδρυματική μέρημνα. Και επιπρόσθετα, η υπηρεσίες κοινότητας ε, δεν ε, ήταν σαφές αν θα προωθούσαν την ε, συμμετοχή των ανθρώπων αυτών, την ένταξη των ατόμων. Επίσης, υπήρχαν λίγες πληροφορίες για την κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία σε αυτές τις συγκεκριμένε χώρες. Αυτή είναι πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί αν δεν έχει υπάρξει ανάλυση των προβλημάτων και των πόσων ανθρώπων είναι σε ιδρύματα τα κενά στις υπηρεσίες που προσφέρονται, τότε θα είναι δύσκολο τα κρατημέλη να σχεδιάσουν πώς θα αντιμετωπίσουν και θα καλύψουν αυτά τα κενά. Έτσι λοιπόν ήταν γλαφυρή η έλλειψη πληροφοριών. Επίσης, είναι ασαφές τι εννοούσαν τα κρατημέλη όταν μιλούσαν για υπηρεσίες ε, κοινωτικέ στη ζωή στην κοινότητα. Και ουσιαστικά κάποια από αυτά τα κονδύλια θα συνεχίζονται να επενδύονται σε ιδρυματική μέρημνα. Αυτή είναι μια σύνοψη των ησυχιών και θα δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφο. Ευχαριστώ. Να συνεχίσω. Η έκθεσή μας τονίζει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ότι ουσιαστικά παρακολουθεί πώς χρησιμοποιείται τα ευρωπαϊκά κονδύλια Μέχρι τώρα ξέρω κάποιες περιπτώσεις ε, που ενημερώθηκε η Κομισιόν για την μη χρηστή χρήση των κονδυλίων. Η κοινωνία των πολιτών έχει διδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Από το 2014 έχουμε ευτυχώς τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεντολογίας ε, ε, για την εταιρική σχέση και λέει ότι θα πρέπει να, συμμετέχουν, να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών σε όλα τα στάδια ε, χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Εδώ βρήκαμε κάποια προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το εξή. Ναι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνική βοήθεια για να οικοδομηθεί η ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να συμμετέχει καλύτερα στις επιτροπές παρακολούθησης. Αν λοιπόν τα κρατημέλη θέλουν να εμπλέξουν την κοινωνία των πολιτών, πρέπει να διασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει μέχρι τώρα. Επίση, χρειαζόμαστε καλύτερο σύστημα παρακολούθηση και σύστημα καταγγελιών στα κρατημέλη Έτσι ώστε να ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία για να καταθέσει κανείς μια καταγγελία, τι συμβαίνει όταν κάποιος καταθέτει μια καταγγελία. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, δεν έχουν συσταθεί αυτά τα συστήματα και η ΝΑΕΛ, δική μου οργάνωση, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για το θέμα αυτό και που λέγεται Ευρωπαϊκά Ταμεία για την πρόθεση των δικαιωμάτων μας. Επίσης, έχουμε μια σύντομη μελέτη εδώ για τη Σλοβακία στην έκθεση. Όπως είπε και η Πρόεδρος, η Επιτροπή Αναφορών επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σλοβακία και τα προβλήματα είναι τα εξή. Δεν είναι η Σλοβακία η μόνη χώρα που έχει τέτοια ζητήματα. Απλώς ε, μας ε, δείχνει ουσιαστικά τα προβλήματα που υπάρχουν στις χώρες ε, όπου δαπανώνται τα κονδύλια. Η δρυματική μέρημνα είναι ένα μοντέλο μερίμνας που κυριαρχεί στη Σλοβακία. Ουσιαστικά βρήκαμε ότι υπάρχουν ε, περίπου 38.900 θέσεις ε, σε ιδρύματα και πάνω από 4.000 ε, παιδιά βρίσκονται σε ιδρύματα. Και από ό,τι φαίνεται δημιουργήθηκαν περαιτέρω 5.000 θέσεις σε ιδρύματα χάρη στην υποστήριξη των διαρθρωτικών τομείων. Εξακολουθεί να υπάρχουν ε, κάποιες ανησυχίες στις Σλοβακίας σε σχέση με τη σημερινή προγραμματική περίοδο. Αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη πολιτικής βούλησης, ε, με το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν συμμετέχει και δεν κατανοεί τη διαδικασία. Υπάρχουν λοιπόν και πάλι καθυστερήσει ε, για το εθνικό πρόγραμμα από ιδρυματικοποίηση, δηλαδή για το πώ θα χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για να προωθηθούν εναλλακτικέ στην ε, ναι, Ιδρυματική μερίμνα. Αυτό τονίστηκε στη μελέτη για τη Σλοβακία που έγινε για την Επίτροπη Αναφορών. Υπήρχε και αυτή η απέτηση τέρη η ΜΚΟ και, μία, και ένα από τα πανεπιστημία θα πρέπει να συγχρηματοδοτήσουν το project από ιδρυματικοποίησης. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι σωστό στη Σλοβακία, όπως ε, και σε πολλές ε, άλλες χώρες, ο τρόπος που χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες ε, ουσιαστικά ενισχύει, την ιδρυματική μέρημνα. Και κάποιος λαμβάνει χρηματοδότηση από τον κεντρικό προϋπολογισμό. αν βρίσκεται σε ιδρυματική μέρημνα, ενώ αν επιλέξει να ζει στην κοινότητα, δεν υπάρχει αυτή η οικονομική αρρωγή. Κάναμε διάφορες συστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βελτιώσει τη συλλογή των δεδομένων. Δεν ε, ήρχε τα τελευταία χρόνια μία πλήρης έκθεση που να εξετάζει το τι γίνεται με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδρύματα. Έχουμε έναν αριθμό 1,2 εκατομμύρια από την έκθεση του 2007. Χρειάζεται επίσης καλύτερη παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε σχέδιο ε, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για ιδρυματική μέρημνα και πρέπει επίσης να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών και να εφαρμοστεί ο κώδικας διοντολογίας για την εταιρική σχέση. Η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στα κράτη-μέλη για το πώς θα εφαρμόσουν καλύτερα τον κώδικα διοντολογίας. Και τέλος, έχουμε κάποιες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Η πρώτη θα ήταν να αναπτύξουμε μια πλήρη στρατηγική για τη μετάβαση από την ιδρυματική μέρημνα στη ζωή στην κοινότητα. Η δεύτερη σύσταση είναι να διασφαλιστεί καλύτερο συντονισμός ε, μεταξύ των μέτρων που υποστηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και ε, από τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλαδή για το πώς γίνεται η στέγαση όταν ε, οι άνθρωποι μετακινούνται από τα ιδρύματα να έχουν και την κατάλληλη υποστήριξη. Η τρίτη σύσταση είναι να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε project ε, ε, χρηματοδοτείται από τα ιδρυτικά ταμεία θα προωθεί και την κοινωνική ένταξη και όχι στο να τοποθετούνται σε μικρότερα ιδρύματα οι άνθρωποι. Πρέπει να επικεντρωθούμε πώς ζουν οι άνθρωποι, στην ε, συμμετοχή του στην κοινωνία, την κοινωνική του ένταξη κτλ. Όχι στα κτίρια. Και επίση να εμπλέξουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, του εμπειρογνώμονε σε διάφορου τομεί και φυσικά να εμπλακούν και ήδη οι άνθρωποι με αναπηρίε στο να αποφασίσουν ποιε υπηρεσίε θα πρέπει να αναπτυχθούν και πώ θέλουν να λάβουν υποστήριξη. Αυτά από εμά. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σα αν έχετε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε καθυστερήσει κάπως, ολοκληρώθηκε το πρώτο πάνελ. Οι τρεις ομιλητές μας έδωσαν πολύ υλικό για την Επιτροπή Αναφορών ως προς τις αναπηρίες σε σχέση με τη συνθήκη του Μαρακές και η Επιτροπή Ρέτζι Επίσης είναι συναρμόδια με την ΠΕΤΗ σε σχέση με την πρώτη εισήγηση για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Και θα δεχτούμε όλες τις ε, υποδείξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στους συμμετέχοντας και η Σολετάτ Καμπεσόν αναλαμβάνει το δεύτερο αυτό πάνελ. Ευχαριστώ Ρώσα, καλημέρα σας. Όπως είπε και η Ρώσα, έχουμε μία μικρή καθυστέρηση, γιατί στη συνέχεια έχουμε να ασχοληθούμε και με αναφορές για αναπηρίες. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρες, μέρος, πάνελ και θα μιλήσουμε για την αναθεώρηση της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες. Η κυρία Ελπίδα Αποστολίδου έχει το λόγο εξ ονόματος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σε αυτό το workshop θα ήθελα να ασχοληθούμε με την εργασία του Ombudsman. Ε, η βασική μας, το βασικό μας μέλημα είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους με αναπτύξεις ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει κακοδιαχείριση από τα ε, θεσμικά όργανα ή τους φορείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οποιοδήποτε ε, έχει την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει αναφορά. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα νομική εκπροσώπηση. Καλύπτουμε πολλά θέματα, δηλαδή προσβασιμότητα σε κτίρια Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσβασιμότητα σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοηματική γλώσσα, χρήση νοηματικής γλώσσας και παραδείγματα επιλογής και εργασίας. Δηλαδή είχαμε έναν υποψήφιο που είχε προβλήματα ακοής γιατί δεν του δόθηκε επιπλέον χρόνος να ανταποκριθεί. Ε, δεν υπήρχε κακοδιαχείριση εδώ γιατί στον, ε, διαγωνισμό έψο είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι προτεραιότητες. Όμως όταν, υπάρχει... όταν υπάρχουν προβλήματα ακοής οι διαγωνισμοί έψω μελλοντικά θα πρέπει να χορηγούν περισσότερο χρόνο σε υποψηφίους με προβλήματα ακοής με βάση τη δήλωση του, των Ηνωμένων Εθνών ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσληψιμότητα ανθρώπων με προβλήματα ακοής, αυτό ήταν μία εύλογη περίπτωση. Είδαμε όμως ότι ο αριθμός ε, αναφορών είναι περιορισμένος. Γι' αυτό θα ήθελα και εσείς να μας χορηγήσετε δεδομένα με τις δικές σας αναφορές. Επίσης, η διαμεσολαβητής θέλει να δει πού υπάρχουν ελλείψεις στα θεσμικά όργανα και θεωρούμε ότι τα δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ σημαντικά γιατί μας δείχνουν πού υπάρχουν ελλείψεις. Ένα από τα θέματα του διαμεσολαβητή αφορά τα θέματα σύνοχης και τη χρήση διαφορετικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων για πολίτες με αναπηρίες. Έτσι γίνεται καλύτερη χρήση των ταμείων. Μία εκπρόσωπος μίλησε για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση σε σχέση με τα ίσα δικαιώματα το Μάιο του 2016. Μετά τα συμπεράσματα και τα σχετικά παράπονα και αναφορές, ο διαμεσολαβητής ξεκίνησε μία έρευνα σε σχέση με το ασφαλιστικό η υπηρεσιακή κατάσταση μιλά για πλήρη επιστροφή ιατρικών εξόδων όταν υπάρχει σοβαρή ασθένεια. Για να θεωρηθεί όμως μια ασθένεια σοβαρή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το θέμα του προσδόκιμου ζωής. Αυτή η ιατρική προσέγγιση όμως δεν λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό μοντέλο όπως δείχνει και η νομολογία του ΔΕΚ. Αυτές οι έννοιες της ασθένειας και των αναπηριών δεν είναι ταυτόσιμες και το ΔΕΚ μίλησε για τον ξεχωριστό τους ε, χαρακτήρα. Το χαμηλότερο προσδόκιμο δεν αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις πολλές αναπηρίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία του ανθρώπου, αλλά δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο ως προς το προσδόκιμο ζωής. Όμως υπάρχουν πολύ υψηλότερα ιατρικά έξοδα και δεν μπορούν τα άτομα αυτά να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή όπως η υγιής. Γι' αυτό ζητήσαμε ειδικά κριτήρια για την κάλυψη ιατρικών εξόδων για πρόσωπα με αναπηρία. Λάβαμε την απάντηση Επιτροπής και την αναλύουμε. Στα πλαίσια αυτά λάβαμε και μία επιστολή από την Επιτροπή Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άτομα με αναπηρία. Ένα άλλο θέμα είναι η προσβασιμότητα στους ιστοτόπους θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και να δούμε κατά πόσο υπάρχει επιγραμμική πρόσβαση. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο υπάρχει ουσιαστική προσβασιμότητα και ε, ως προς τη νοηματική και τη γραφή μπράγη για όσους εργάζονται στη, στους ιστοτόπους. Η Επιτροπή είπε ότι οι πληροφορίες στη ε, νοηματική κινείται πέρα από το επίπεδο συμμόρφωσης με βάση τον κώδικα προσβασιμότητας 2. Η αποτίμηση προσβασιμότητας λαμβάνει υπόψη της επικαιροποίησης. Και ως προς την κατάρτιση η Επιτροπή είπε ότι προβάλλει ένα μάθημα προσβασιμότητας, μια ειδική κατάρτιση. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η διαμεσολαβητή σε επόμενη φάση και θα λάβουμε υπόψη τις ε, πρόσφατες ε, εξελίξεις, ιδιαίτερα την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους και σε δημόσιους φορείς. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κανόνες προσβασιμότητας και θα πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουν τα θεσμικά όργανα στο μέλλον. Σε σχέση με το δικό μας ε, website θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει πιο φιλικό προς το χρήστη και πιο εύκολα προσβάσιμο. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να προβληθούν καταγγελίες σε 24 γλώσσες. Τώρα ε, έχουμε και μία εξωτερική αποτίμηση και αξιολόγηση του ιστοτόπου του διαμεσολαβητή. Επίσης, μέσα στα πλαίσια του πλαισίου εποπτείας θα προβάλλουμε ε, καταγγελίες έτσι ώστε να υπάρξει πλήρη χρήση της σύμβασης. Θα θέλαμε λοιπόν όλο το χρήσιμο input για να φτάσουμε σε έναν μετρήσιμο αντίκτυπο όλων αυτών των μέτρων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ στη συνέχεια από την Επιτροπή δικαιωμάτων των δύο φίλων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κυρία Μάρθα Στίκινγκς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση να πάρω το λόγο στη σημερινή συνάντηση. Να συγχαρώ την Επιτροπή για το γεγονός ότι έχει συστηματοποιήσει τέτοιου είδους συναντήσεις και εκδηλώσεις και το γεγονός ότι εξετάζουμε ιδιαίτερα τα θέματα ατόμων με αναπηρία. Αυτό δεν ευαισθητοποιεί ιδιαίτερως για τα θέματα αυτά και για τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατομών με αναπηρία του ΟΗΕ. Και χαίρομαι που καταφέραμε να συμβάλλουμε όχι μόνο με την παρουσία μας, αλλά και με την παροχή ε, στοιχείων και δεδομένων από τις αναλύσεις μας. Και σήμερα τονίζονται δύο βασικοί ρόλοι που θα μπορούσε να δραματίσει η Επιτροπή Αναφορών σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Και αυτό ασφαλώς αφορά και το ρόλο που μπορούν να παίξουν και άλλα όργανα σε ό,τι αφορά την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Καταρχάς, οι μεμονωμένες ε, ε, ενστάσεις και περιπτώσεις και αγωγές στα πλαίσια και της σύμβασης και των γενικότερων νομικών πλαισίων. Ένα δεύτερο θέμα αφορά και πιο διαρθωτικά ζητήματα. Πέρα από τις μεμονωμένες, μεμονωμένα προβλήματα, κάποιες οριζόντιες προκλήσεις που αντιμετωπίζεται σε ό,τι αφορά α, ε, τη σωστή διαμορφώση του δικαίου. Και ασφαλώς και τα δύο αυτά στοιχεία έχουν σημαντικό ρόλο να διαρματίσουν σε ό,τι αφορά την προστασία και το ρόλο προστασίας των εκστρατιών, των μηχανισμών προστασίας στα πλαίσια τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με την Απειρία, του ΟΗΕ, αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση Κουσιαστικών Συνθήκων. Η Υπηρεσία Θεμελιδιών Δικαιωμάτων ασφαλώ δεν έχει εντολή να αντιμετωπίζει και να διεκπαιρεώνει τέτοιε ενστάσει. Ε, δεν είμαστε δικαστικό σώμα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εργασία μας, είναι σημαντικό τέτοιες ενστάσεις και αναφορές να μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία, τοποθετήσεις, συστάσεις εμπερογνωμόνων, προκειμένου να είναι σωστά τοποθετημένες και να έχουν σωστή τεκμηρίωση, κατανοώντας σε βάθος την κατάσταση. Και θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τρεις τρόπους με τους οποίους η Υπηρεσία Θεμελιδών Δικαιωμάτων ως κέντρο αριστείας για τα δικαιώματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει στοιχεία στην Επιτροπή Αναφορών και να βοηθήσει το μηχανισμό για την υποβολή ενστάσεων. Καταρχάς, τι κάνουμε, ένας πρώτος ρόλος είναι η συλλογή στοιχείων και τεκμηρίων ανάλυση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μέσω των θεματικών μας εκθέσεων για την ψηφιακή συμμετοχή, βία κατά των παιδιών με αναπηρία, οποιαδήποτε θέμα για να αφορούν. Μέσω λοιπόν των δεδομένων αυτών και των αναλύσεων μπορούμε να δούμε ποιο είναι το κενό και το χάσμα στην εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως τη ζει το άτομο με την αναπηρία. Πέρα από τις θεματικές αυτές έρευνες, κάνουμε και πάρα πολλή δουλειά για να βρούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ποια είναι η πρόοδος και οι τάσεις ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της σύμβασης και εστιαζόμαστε ιδιαίτερα στο θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια μέσω ενό ιδιαίτερου κεφαλαίου στην ετήσια έκθεσή μα, το οποίο εξετάζει ακριβώ την εφαρμογή του CRPD, τη Σύμβαση για Δικαίωμα των Ατόμων Αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δημοσιευτεί του χρόνου και ένα δεύτερο τμήμα στο κεφάλαιο αυτό. Εδώ λοιπόν εντοπίζονται κάποιοι από του κοινού τομεί όπου γίνονται αλλαγέ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της σύμβασης και επίσης εξετάζουμε πώς ε, εφαρμόζονται τα μέτρα για να καταπολεμήσουν τις διακριτικές μεταχειρήσεις κατά των ατόμων με αναπηρία. Και αυτό εντάσσεται και στη γενικότερη εργασία μας, όπου εξετάζουμε την αναπηρία πιο οριζοντία και το πιο θα πρέπει να είναι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να δράσουμε. Εξετάζουμε επίσης το πώς ε, τα κρατημέλη εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού για τα διευθυντικά ταμεία. Για παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια είδαμε πώς εφαρμόζονται τα ταμεία διευθυντικής ανάπτυξης και σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία και σε αυτό θα επανέλθουμε σίγουρα σε δύο χρόνια ε, γιατί αρχίζουν να εφαρμόζονται τα διευθυντικά ταμεία σε ό,τι αφορά την τρέχουσα πραγματική περίοδο. Κατά δεύτερον, ένα άλλο τρόπο ε, με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε την Επιτροπή Αναφορών είναι με την ανάπτυξη των δικτών ανθρωπινών δικαιωμάτων, γιατί αυτό το ξέρετε πολλοί από εσά. Υπάρχουν ήδη εφαρμοσμένοι δείκτε για τα 28 κρατημέλη βάσει του άρθρου 29 τη σύμβαση, δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή. Και επίση έχουμε αναπτύξει μια σειρά δικτών για το άρθρο 19 τη σύμβαση. Ε, το ακούσαμε σήμερα το πρωί αυτό Συλλέγουμε λοιπόν δεδομένα και από τα 28 κρατημέλη για να καταρτήσουμε τους δείκτες αυτούς, τους οποίους και καταρτίζουμε στην παρούσα φάση. Με χαρά διαπιστώνω ότι πολλούς από τους δείκτες που αναπτύσσουμε αντικατοπτρίζουν τα θέματα τα οποία ανακύπτουν και στην έκθεση τα οποία παρουσιάστηκαν και σήμερα άλλωστε αποτυπώνουν για παράδειγμα το θέμα της προσβασιμότητας στις, στις ε, υπηρεσίες υποστήριξης. Έχουμε λοιπόν τη νομική υποχρέωση παροχής πρόσβασης ε, σε τέτοια συστήματα πληροφόρησης. Κοιτάμε που υπάρχει σχετική χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά πόσον αυξάνεται ή μειώνεται αυτή η χρηματοδότηση με την πάρδα του χρόνου. Και επίσης εξετάζουμε πόσα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές. Εδώ ασφαλώς έχουμε ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο, το οποίο και πάλι το ακούσαμε και σήμερα το πρωί, η έλλειψη συστηματικών και εντελεχών στοιχείων, τα οποία θα μας επέτρεπαν να εφαρμόσουμε με κάποιο σωστό τρόπο και σκόπιμο τρόπο τους δείκτες αυτούς για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, βλέπουμε πόσο ο ΦΡΑ μπορεί να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω σε ό,τι αφορά το μηχανισμό για την υποβολή τέτοιων ε, παραπώνων και ενστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα εργαλείο clarity, σαφήνειας. Ε, είναι λοιπόν ένα εργαλείο αυτό το οποίο διατίθεται στο δίκτυο, είναι προσβάσιμο και κατέστηται όλο και πιο προσβάσιμο να σας πω οι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν εδώ να δουν ποιος είναι ο πιο ε, άμεσος και σχετικός ε, μηχανισμός υποβολής ενστάσεων που θα μπορούσε να ταιριάξει στην περίπτωσή τους. Καλύπτει 15 κρατημέλη στην παρούσα φάση και θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιείται για να εντοπίζονται οι υπηρεσίες για την ισή μεταχείριση, οι οργανισμοί, οι διαμεσολαβητές, για να μπορεί ο καθένας να δει σε ποιον τέτοιο μηχανισμό θα έπρεπε και θα μπορούσε να απευθυνθεί. Γιατί συχνά ξέρετε υπάρχει μεγάλη σύγχυση για το ποιο είναι το πιο σωστό και αρμόζον σώμα στο οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί κανείς. Θα ήθελα κλείνοντα να αναφέρω δύο τομείς ε, στους οποίους η εργασία του Οργανισμού Ανθαμελιδών Δικαιωμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με αυτά που ακούσαμε και σήμερα το πρωί. Το πρώτο αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπε και ο Μάρκ προηγουμένω, στι αρχέ του έτου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μια επίσημη νομική τοποθέτηση τη υπηρεσία μα σε ό,τι αφορά το άρθρο 33.2 τη Σύμβαση για τη Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε ό,τι αφορά το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην εκνομοδότηση λοιπόν αυτή, εξετάσαμε διάφορα ζητήματα τα οποία από τη σύσταση, τη εντολή, Τη λειτουργία του πλαισίου και ακούσαμε διάφορε απόψει ασφαλώ για το πώ μπορεί να βελτιωθούν οι υφιστάμενε δομέ και πώ μπορούν να ενισχυθούν και σε βάθο χρόνου. Ένα τέτοιο θέμα ήταν να εξετάσουμε τα καθήκοντα του πλαισίου. Και είδαμε ότι η Επιτροπή του CRPD της ε, Σύμβασης για τα των Ανθρώπων με την Αναπηρία ε, έχει κάνει διάφορες συστάσεις και συμφωνούμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, τη συλλογή στοιχείων κτλ. Φυσικά, οι ρόλοι αυτοί σε μεγάλο βαθμό εκτελούνται και από τα μέλη του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρούμε ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω μια νομικά δεσμευτική πράξη που θα αποτελεί βάση για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης μέσω προβλέψης δυνατότητας ε, γνωμοδότησης ε, με ίδια πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι το Κοινοβούλιο με τα άλλα θεσμικά όργανα ήδη έχει δυνατότητα να ζητά την επίσημη νομική τοποθέτηση του ΦΡΑΚ. Τους καλούμε να το κάνουμε αυτό που το επιθυμούν και που τα χρειάζονται. Σε ό,τι αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση και την ε, μετάβαση από τη δραματοποίηση σε μια ανεξάρτητη ζωή με κοινωνική υποστήριξη. Σε πέντε καθημέρι λοιπόν κοιτάμε τα θέματα, ένα από τα οποία είναι και η Σλοβακία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που κάποια από τα πρώτα πορίσματα α, της ε, έρευνας μας αυτής υποστηρίζουν τη διερευνητική αποστολή. Τα Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τη Βουλγαρία, τη Φιλανδία, την Ιρλανδία και την Ιταλία και τη Σλοβακία Ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν να βρούμε κάποια από τα βασικά, τους βασικούς δείκτες, κάποιους από τις βασικές δείκτες που οδηγούν ή απομακρύνουν από την ιδρυματοποίηση. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε σε συνδυασμό και με τις προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και πορίσματα σε ό,τι αφορά και το άρθρο 19 για την απομάκρυνση από την δραματοποίηση. Αυτά. Και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, εφόσον επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τι Αναπηρίε, η κυρία Κάθριν Νιούτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο και ευχαριστώ και την Επιτροπή Αναφορών για την πρόσκληση. Θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ την εκτίμησή μου όπως η Μάρθα από το ΦΡΑ που η Επιτροπή Αναφορών έχει μια συστηματική προσέγγιση σε σχέση με το ρόλο της απέναντι στα άτομα με Ευχαριστώ και την συνεχή σας δέσμευση για το θέμα της σύμβασης του Μαρακές. Εμείς πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα το διεκπαιρεώσει αποτελεσματικά αυτό το θέμα και θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τα εμπόδια που υπάρχουν με τα κράτη-μέλη για να γίνει πραγματικότητα η Σύμβαση του Μαρακέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, να συνεχιστεί και η πίεση σε ό,τι αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά τριφθετικά ταμεία. Θε, το να ακούμε ότι χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια για να δημιουργούνται νέες θέσεις ε, σε ιδρύματα είναι λυπηρό. Νομίζω ότι όλοι σήμερα είμαστε συγκινημένοι. Ξέρουμε ότι οι πολιτικοί θεσμοί στην Ευρώπη, στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που αναμένουν οι άνθρωποι, οι πολίτες. Ξέρουμε ότι εργαζόμαστε για να προωθήσουμε και τα δικαιώματα των ανθρώπων ευηρίες, αλλά και τη λογοδοσία των θεσμών προς τους πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ενθαρρύνω την Επιτροπή Αναφορών ε, να παρακολουθεί τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για να είναι σίγουροι ότι πραγματικά θα εξακολουθούν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ανθρώπων με αναπηρία. Εμείς, αν δεν μας γνωρίζετε, είμαστε μια οργάνωση ομπρέλα και εκπροσωπούμε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη Δημιουργηθήκαμε πριν 20 χρόνια περίπου για να προωθήσουμε τα δικαιώματα των ατόμων με εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμαστε με το ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σύνεψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανεπηρίες ε, και κλείνει τα δεκαέτη η σύμβαση αυτή φέτος ήμασταν ενεργοί στη διαδικασία αναθεώρησης μαζί και με τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Αναφορών και συνεργαζόμαστε και εργαζόμαστε συστηματικά για να υπάρχει follow-up ε, των διάφορων συστάσεων της Επιτροπής. Είμαστε ικανοποιημένοι που εκδόθηκε πέρσι η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και μαζί με το European Disability Intergroup διερευνούμε τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν για την υιοθέτηση της σύμβασης και φυσικά θα συνεχίσουμε να δίνουμε σύμβαση στην Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας. Τώρα, ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση των συστάσεων είχαμε μια συνάντηση προκειμένου να μπορέσουν και οι stakeholders να δώσουν τη δική τους συνεισφορά για τις συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για θέματα που θεωρούν να είναι ζωτικά. Μιλήσαμε για τα τρία επίγοντα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και θέματα που θεωρούνται επίγοντα από όλου του προκεκλημένου, στο να υπάρχει πλήρη υποβολή έκθεση γι' αυτό και μέχρι τα τέλη του έτου. Η διαδικασία λοιπόν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Υπό την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσει feedback στην Επιτροπή για τα τρία σημαντικά θέματα και εμείς θα δώσουμε κατόπιν feedback ε, στην Επιτροπή κατόπιν ενό έτου. Αυτό θα γίνει φέτο. Επίσης εξετάσαμε τις διάφορες ε, συστάσεις ε, που απευθύνονταν σε διάφορες διευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συναντηθήκαμε με διάφορους επιτρόπους και με άτομα που εργάζονται στι υπηρεσίες για το πώς θα προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Βλέπουμε πολλές ευκαιρίες όπως ε, στο να δίνουμε, να προωθούμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, να προωθούμε τα δικαιώματα των ατόμων εμπειρία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών και στην Πρατισλάβα. Αυτό το επόμενο, το επόμενο Σαββατοκυριακό θα έχουμε μία διάσκεψη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, της Σλοβακικής Προεδρίας και θα εξετάσουμε τη διαδικασία της παρακολούθησης και της συνέχισης των συμπερασμάτων στα οποία καταλήξαμε. Συνεργαζόμαστε μαζί με τα μέλη μας για να υποστηρίξουμε την Επιτροπή της Γενέβης. Δηλαδή πώς θα γίνει η προετοιμασία των εκθέσεων του Πικοδημητικού διαλόγου, αλλά για πρώτη φορά το Σάββατο θα δούμε τι ακριβώς κάνει κανείς όταν λάβει τις συστάσεις. Δηλαδή, ποιε είναι οι πιο επιτυχείς δράσεις για να διασφαλίσουμε ότι θα φέρουν πραγματική αλλαγή στι συστάσεις αυτέ σε χώριο επίπεδο. Μια άλλη νέα δράση από το EDF ως προς το ρόλο μας εντός του πλαισίου είναι το εξής. Θα υλοποιήσουμε μια σειρά εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη θα είναι έτοιμη για τα τέλη Νοεμβρίου. Στις 29 και 30 Νοεμβρίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα άτομα με Τι θα κάνουμε με αυτή τη σειρά θα εξετάσουμε διάφορα σημαντικά θέματα και θα δούμε ποιε είναι οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωση και κρατών μελών. Πρώτη έκθεση που ελπίζουμε θα την έχουμε στα χέρια μα την επόμενη εβδομάδα, απλώ θα θέσει το σκηνικό. Έχουμε τη δέκατη επέτειο τη σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατομών Επηρείας, να δούμε τι συμβαίνει εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε τη κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου, ποιε χώρες έχουν κάνει δηλώσεις που ουσιαστικά δεν σέβονται τις προθέσεις της σύμβασης και το πνεύμα της σύμβασης και θα τονίσουμε τις διάφορες προκλήσεις. Κατόπιν, τα επόμενα έτη, θα αντιμετωπίσουμε άλλα συγκεκριμένα ζητήματα και άρθρα για να ενθαρρύνουμε να γίνει κάποια σύγκριση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη το κάνουμε αυτό στις συναντήσεις του Συμβουλίου μας και στις Γενικές Συνελεύσεις. Δηλαδή εξετάζουμε πώς δρούν τα κρατημέλη, αλλά θέλουμε να το συστηματοκοποιήσουμε Ουσιαστικά είναι μια σειρά που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία λοιπόν από την πλευρά μας ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης. Πρόσφατα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επισκεφτήκαμε την Ελλάδα για να δούμε τι γίνεται με τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες με αναπηρίες. Ε, η Ελλάδα πριν ήταν χώρα διέλευσης, ενώ τώρα έχει γίνει χώρα προορισμού. Και πάρα πολλοί ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, ασυνόδευτοι ενήλικοι, άνθρωποι με αναπηρίες έχουν παραμείνει στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν μαζί με την ΟΚΕ στις 14 Φεβρουαρίου θα κάνουμε μια σχετική ακρόαση για να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δράσεις της για να διασφαλίσει ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των προσφύγων με αναπηρίες. Θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Επιτροπή στην Εμμανουέλ Γκράνς για να μας μιλήσει για το πώς ε, έχει ε, ενημερωθεί η πολιτική Εμείς ε, δεν συμμετέχουμε επίσημα στη σύμβαση, γι' αυτό κάθομαι και σε αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτό του workshop και για την υποστήριξη της Επιτροπής ΠΕΤΗ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη των ε, πολιτών με αναπηρίες που, ε, στους οποίους μάλλον επενδύουμε πολύ πολλά αναφέρθηκαν σήμερα το πρωί που θα ήθελα να συζητήσω, αλλά δεν θέλω να σας απασχολήσω για 20 λεπτά. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Ε, έγινε λόγος για την απόσυρση της Κομισιόν από την επίσημη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και όπως σας είπα ε, και όπως είπα και στην ΕΟΚΕ η Επιτροπή δεν αποσύρεται από τέτοιες διαδικασίες. Γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολο να βρούμε τη σωστή διαδικασία να εξηγήσουμε τι έπρεπε να γίνει σε σχέση με το 2012 που δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο και να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από νομικής πλευράς. Χτες ε, είχαμε την επιβεβαίωση της διαδικασίας της ε, επωνομαζόμενης Fish Grease έτσι ώστε να επισημοποιήσουμε αυτή την απόσυρση από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ένα non-paper, για ένα άτυπο έγγραφο σε σχέση με τη διαδικασία του 2012 για να δείξουμε ε, τι θα ισχύσει σε αυτό το πλαίσιο χωρίς την Κομισιόν. Πρόκειτο για το πλαίσιο εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι μια πιο μακροχρόνια ε, διαδικασία που αφορά και το πλαίσιο και τα θεσμικά όργανα. Αυτό το θέμα δεν το θίξαμε και θεωρούμε ότι η επίσημη απόσυρση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα γίνει σύντομα μέχρι το τέλος του έτους. Θα διευθετηθεί το όλο ζήτημα και έτσι θα έχει και νομική υπόσταση αυτή η απόσυρση. Αυτό δεν αλλάζει τα σημεία εστίασης για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι είτε για την προώθηση και την εποπτεία της σύμβασης ε, μέσα στην οποία δρούμε με τους ε, πόρους που διαθέτουμε σε αυτούς τους τομείς και για να υποστηρίξουμε και τις ΜΚΟ που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα κάθε χρόνο ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με τις ε, ΜΚΟ έτσι ώστε να έχουμε ένα σκόπιμο feedback. Αυτό ακριβώς ε, μας ε, απασχολεί και το οποίο ήδη εκφράσαμε και που έχει σχέση και με τη σύνταξη των εγγράφων μας και την διάρθρωση της πολιτικής μας. Πρόκειται για βέλτιστες πρακτικές και για ανταλλαγή αυτών. Θέλουμε να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση για τη σύμβαση. Χαιρόμαστε για το ότι πρέπει να αναλάβουμε πολλές δραστηριότητες και για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή απόψεων για την επιτόπια δράση μας. Εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και μαζί για τις, ως προς τις σας αναφορές και τις καταγγελίες που λαμβάνουμε εμείς. Ε, είναι ε, δύσκολο να τις διαχειριστούμε πάντα αυτές τις καταγγελίες γιατί δεν άπτονται θεμάτων αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για θέματα που πρέπει να επιληθούν και σε κρατικό επίπεδο, είτε πρόκειται για τα επιδόματα αναπηρίας ή τις καθημερινές διακρίσεις και δυστυχώς δυστυχώς δεν είναι τομείς στις οποίους ε, έχουμε, για τις οποίους έχουμε αρμοδιότητες. Αποτελούν όμως ένδειξη ε, της όλης μας συλλογιστικής και που θα πρέπει να τύχει ανάλυσης ε, πιο ολοκληρωμένα. Εντάχει λοιπόν θα ήθελα να σας πληροφορήσω ως προς την εποπτεία της σύμβασης ότι αυτή τη βδομάδα θα αρχίσει η ενδοϊπηρεσιακή διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Αναπηριών και αν όλα πάνε καλά με τις διαβουλεύσεις θα έχουμε το έγγραφο στις αρχές Δεκεμβρίου κάναμε μία αποτίμηση της κατάστασης σε σχέση με τη στρατηγική για τις αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσετε και εσείς να ανταποκριθείτε στην ανάλυση της κατάστασης. Ως προς τα διαρθρωτικά ταμεία, Εκφράστηκαν πολλές σχέσεις, το θέμα είναι ζωτικής σημασίας μέσα στα πλαίσια των ε, θεσμικών λειτουργιών. Έχουμε μία περίοδο προγραμματισμού η οποία δεν είναι τάχιστη και έχουμε ε, φυσικά μία ε, από κοινού διαχείριση με τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη αυτή τη συνεργασία. Υπάρχει μία θεσμική λειτουργία, αλλά θα θέλαμε τη συνεργασία τους. Χρειάζεται μία διαδικασία εποπτείας και από την κοινωνία των πολιτών, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το θεσμικό αυτό όργανο που αποτελεί σύνδοσμο με τα κράτη-μέλη. Και είδαμε μεγάλη ικανοποίηση, μια πραγματική συνένεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει λοιπόν ε, ένας θα μπορούσα να πω σαν ημάντας διαβίβασης της κίνησης αυτής. Υπάρχει λοιπόν ευαισθητοποίηση και στις ε, υπηρεσίες της Επιτροπής για να υπάρξει χρηστή εφαρμογή και χρήση γενικότερα των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Ε, υπολείπεται όμως πολλή εργασία. Πρέπει να αλλάξουμε τις πρακτικές που υφίστανται για να γίνουν χρηστότερες και από το ε, Κοινοβούλιο, ΦΡΑ και μη κυβερνητικέ. Όμως ε, μας απασχολεί αυτό το ζήτημα, γίνονται συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους εμπειρογνώμονες και είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να συνεργαζόμαστε για να έχουμε ε, μία διαδικασία σωστής εποπτείας. Ελπίζω να σας έδωσα ορισμένα στοιχεία πληροφόρησης άκρος ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Και τέλος, όπως είχα πει, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα χρόνου. Και πρέπει φυσικά να ακούσουμε τους αναφέροντες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και Απλώ να σας πω ότι εμεί ω Επιτροπή Αναφορών συνεχίζουμε τι δεσμεύσει μας ε, να έχουμε ουσιαστικά στο στόχαστρο αυτή την προβληματική για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ανάγκες των πολιτών. Ε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ε, σε αυτό, κατά τη διάρκεια του χρόνου για αυτό το θέμα, αλλά φυσικά θα συζητήσουμε και σε άλλα βήματα. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορεί να υπάρχει συζήτηση, αλλά όπως σας είπα πρέπει να δώσουμε το λόγο στους αναφέροντες. Thank you all. Thanks to the panelists. Thanks to the... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Ευχαριστώ και την Αντιπρόεδρο για την ε, συνεδρίαση αυτή. Νομίζω τώρα ότι χωρί χρονοτριβή θα πρέπει να περάσουμε στι συγκεκριμένε αιτήσει. Συγγνώμη, συγκεκριμένε αναφορέ που έχουμε σήμερα. Πρόκειται καταρχήν για την αναφορά 1140 εκ μέρου ε, τη European Guide Dog Federation και τη Assistance Dogs Europe σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβαση ατόμων που έχουν ανάγκη σκύλων βοηθεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον αναφέροντα Παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που εξετάζετε αυτή την αναφορά και που με ακούτε τώρα. Ο David Adams και εγώ ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας ε, πείσουμε μέσω της αναφοράς μας για την ανάγκη Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ή κατευθυντήριων γραμμών σε ό,τι αφορά τη δημόσια πρόσβαση για τους σκύλους βοηθείας ε, ε, και τους χειριτές τους. Ε, φανταστείτε να είστε άτομο με αναπηρία, παραδείγματο χάρη τυφλός ε, ή σε αναπηρική καρέκλα ή να υποφέρετε από επιληψία, από κρίση επιληψίας. Έχετε σχεδιάσει και ανυπομονείτε να βγείτε ένα βράδυ έξω με τους φίλους σας φυσικά, παίρνετε και το σκύλο βοηθεία σας μαζί σας καταρχήν, επισκέφτεστε μια pub, σας επιτρέπουν να μπείτε, αλλά μόνο επειδή ξοδεύετε χρήματα αλλά σας κάνουν και ένα σχόλιο για την παρουσία του σκύλου. Φανταστείτε πώς θα νιώθατε. Και η ιστορία συνεχίζεται. Αφού φύγετε από την ΠΑΚ, σε ένα εστιατόριο, πριν μπορείτε να μπείτε, σας μπλοκάρουν την είσοδο, σας μπλοκάρει την είσοδο διοκτήτη και δεν σας αφήνει να μπείτε λόγω του σκύλου. Φαντάζεστε πώς θα νιώθετε. Αυτά που περιγράφω εδώ δεν είναι κάτι που συμβαίνει περιστασιακά, είναι πραγματική ζωή για οποιοδήποτε διοκτήτη βοηθείας. Εγώ ως ε, μέλος ε, της Assistance Dog Guru έχω ε, ουσιαστικά καταγράψει θέματα πρόσβασης από το 2009 το 2013. Ενενώσαμε τις συνάμε μας με τον David Adams και το European Guide Dog Federation σε ό,τι αφορά τα θέματα δημόσιας πρόσβασης. Είδαμε ότι τα προβλήματα πρόσβασης για τους σκύλους βοηθείας δεν περιορίζονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο. Ανακαλύψαμε ότι το να ταξιδεύει κανείς στην Ευρώπη να επισκέφτεται το τοπικό παντοπολείο δεν είναι πάντοτε μια ευχάριστη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ο οποίο και ο ίδιος χρησιμοποιεί σκύλο και είναι πρόεδρος του EGDF, συνάντησε πολλά προβλήματα πέρσι. Παραδείγματο χάρη, του αρνήθηκαν πρόσβαση αν και ήταν εντάξει όλα του τα χαρτιά σε ένα αεροπλάνο που πετούσε από το Λονδίνο στη Σλοβενία, όπου ο Ντέβιτ είχε οργανώσει μια διάσκεψη της e GDF και έφτασε μια μέρα αργότερα στη δική του διάσκεψη. Ένα άλλο παράδειγμα, του αρνήθηκαν εδώ στις Βρυξέλλες να του δώσουν δωμάτιο στο ξενοδοχείο λόγω του σκύλου του. Ένα άλλο παράδειγμα, ένας οδηγός ταξί, μάλλον οδηγεί ταξί σε όλη την Ευρώπη, ε, και κάποιος οδηγός ταξί δεν ήθελε να πάει τον Ντέιβιτ ε, στο προορισμό του. Στη Γαλλία συνέβη αυτό. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά καταλαβαίνω ότι πήρατε το μήνυμα. Όλα τα προβλήματα προέκυψαν από την παρουσία του σκύλου και τελικά κάτι που θα έπρεπε να έχει ευτυχή έκβαση έγινε φιάλτης. Το να μην είναι κανείς σε θέση να κάνει αυτό που θέλει όταν θέλει να το κάνει, δεν σέβεται τη σύμβαση του ΟΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Καθώς από τότε που κύρωσε τη Σύμβαση Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χρήστε των σκύλων βοηθεία θα μπορούσαν να περιμένουν κάποια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ουσιαστικά αξιώνονται στα δικαιώματά τους για δημόσια πρόσβαση και προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους όπως θα ήθελαν. Ελπίζω να μπορώ να σας πείσω για την ανάγκη Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε κατευθυντήρων γραμμών σε ό,τι αφορά τη δημόσια πρόσβαση για τους κύλους βοηθείας. Σας διαβεβαιώ ότι κάθε ιδιοκτήτης κύλου βοηθείας θα σας ευγνωμονεί αν εκπονήσετε αυτή τη νομοθεσία της κατευθυντήριας γραμμές για να διευκολύνετε τη ζωή τους. Όχι μόνο εκεί που ζουν τοπικά αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Πράττοντας κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στο στρατηγικό στόχο του 2020. Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα για τα άτομα με αναπηρία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και χρειάζεται να σας πω ότι το πάθος και η συμπόνια από πλευρά της Επιτροπής μας παραμένει στο πλευρέ σας και καταλαβαίνουμε πραγματικά τα προβλήματα που περιγράφετε. Πραγματικά σημαίνουν πάρα πολλά αυτά για μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να δώσω το λόγο λοιπόν γρήγορα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Γκριόνς νομίζω είναι η αρμόδια που θα πάρει το λόγο. Δεν ξέρω ποια είναι η υπεύθυνη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι και εμείς ε, έχουμε να εκφράσουμε την συμπόνια μας και συμπάσχουμε με τον αναφέροντα ότι αφορά την κατάσταση αυτή και όλοι έχουμε τέτοιε καταστάσεις στην καθημερινή μας ζωή. Και σε πολλές περιπτώσεις ε, νομίζω ότι αυτό ε, αποδεικνύει ότι υπάρχει άγνοια ουσιαστικά, όχι τόσο πολύ ανοησία, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια διακριτική μεταχείριση που δεν έχει βάση ουσιαστικά σε καμία νομοθεσία. Δεν υπάρχει τυπικά και επίσημα πουθενά γραμμένο ότι οι σκύλοι βοηθείας απαγορεύονται στο τάδε, στο δυναμέρος. Δυστυχώ πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση οδηγία για την ε, καταπολέμηση της διακριτική μεταχείριση το 2008. Βρίσκεται ακόμα στη φάση συζήτηση ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου παρά το γεγονό ότι έχει περάσει πολλή χρόνο. Ελπίζουμε να είναι φετική έκβαση κάποια στιγμή. Και το θέμα αυτό είναι ένα θέμα διακριτικής μεταχείρισης κατά των ατόμων με αναπηρία, το οποίο θα επέτρεπε μια πιο σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στην παρούσα φάση, πέρα από αυτά που έχουν προταθεί. Ελπίζουμε ότι η πρόταση αυτή κάποια στιγμή θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Εμείς εμείς σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα να ανοίξει η συζήτηση. Παρακαλώ, δεν ξέρω συνάδελφοι ποιος θέλει να πάρει πρώτο το λόγο. Κανείς? Μάλιστα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο και πάλι στον αναφέροντα. Α, ο κύριος Πίτερ Γιάρ θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, να μην πειράξω κανένα μικρόφωνο και κάνω και μια ζημιά. Φαντάζομαι ότι όλοι οι συνάδελφοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη σκέψη τους, γιατί η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας άφησε και λίγο άναυτους. Χρειάστηκε να τη σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Εμείς διαπιστώνουμε ότι είναι απλά απαράδεκτη κατάσταση, μη ικανοποιητική, είτε πρόκειται για διακριτική μεταχείριση, όπως και να έχει χρειάζεται μία ρύθμιση. Άρα έχω να ρωτήσω το εξή. Αφελώ πώ, τι είδου ε, νομοθεσία θα χρειαζόταν η οποία θα έκανε, θα έβγαζε νόημα και θα έλυνε τα προβλήματα στην πράξη. Αυτό λοιπόν το ρωτώ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό θα καθορίσει και την υπόλοιπη δραστηριότητά μα. Και προφανώ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Θα πρέπει ενδεχομένω να συμμετέχουν και άλλε ε, αρμόδιες επιτροπές, συναρμόδιες επιτροπές για να ξέρουμε τι συμφέροντα παίζονται. Ήταν ε, μη ικανοποιητική η απάντηση, θεωρώ. Δηλαδή, από τη μία όλα έχουν καλώς, αλλά από την άλλη είναι παραδεκτή κατάσταση. Τι θα πρέπει λοιπόν να γίνει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρο. Άλλος κανείς. Όχι. Μάλιστα. Να δώσω λοιπόν και πάλι το λόγο στον κύριο Φανχέλτερ για να απαντήσει ενδεχομένω αν το επιθυμεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τον συνάδελφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να μας δώσει κατευθυντήρες γραμμές, η νομοθεσία Παρ' όλα αυτά όμω θεωρώ ότι το θέμα δεν πρόκειται ποτέ να επιληθεί. Αν ο κόσμο σήμερα, ενέτη 2016, που μπορεί να ταξιδεύει χωρί περιορισμού στην Ευρώπη, σε αυτό που αποκαλούμε όλοι μία ενιαία Ευρώπη, είναι γελίο αυτό που συμβαίνει. Ναι, καταλαβαίνω ότι από τι χώρε εξαρτάται το κατά πόσο θα κάνουν κάτι ή όχι, αλλά εκεί ακριβώ βρίσκεται το πρόβλημα δεν υπάρχουν αρκετές χώρες που να θέλουν κάτι να κάνουν. Το Βέλγιο, για παράδειγμα. Εγώ εργάζομαι από το 2009 επί της σχετικής νομοθεσίας στο Βέλγιο. Τον Ιανουάριο του 2014 επιτέλους στο φλαμανδικό τμήμα της χώρας εγκρίθηκε η σχετική νομοθεσία το Βέλγιο είναι μικροσκοπικό σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και υπάρχουν τρεις διαφορετικές νομοθεσίες που διέπουν το Βέλγιο. Δεν μπορώ να πάρω το σκύλο μου και να ταξιδέψω από τη Φλάντρα στο γαλόφωνο κομμάτι, γιατί στο γαλόφωνο κομμάτι δεν επιτρέπεται να μπει ο σκύλος. Είναι πραγματικά γελίο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σηκώνει το χέρι ψηλά και λέει «Α, τι θα κάνουμε κι εμείς, δεν φταίμε εμείς». Μα ποιο φταίει τελικά. Η Ευρώπη δεν είναι αυτή που πρέπει να δώσει τις κατευθυντήριε γραμμέ. να νομοθετήσει. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα πρέπει όλοι, μάλλον όλοι έχουν υπογράψει τη συνθήκη αυτή. Και τώρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε δεν είναι δικό μα πρόβλημα. Όταν μίλησα στον Πρωθυπουργό πριν από κάποια χρόνια, τι μου είπε το περιφερειακό φλαμαντικό πρόβλημα δεν μας αφορά. Δεν μπορούμε να δράσουμε. Όταν ήρθα σε επαφή με την οργάνωση Ούνια, όπου μπορεί κανείς να υποβάλει ενστάσεις σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης. Όταν επικοινωνήσα λοιπόν μαζί τους, Αυτό που μου απάντησαν ήταν ότι εμείς προσυπογράψαμε τη σύμβαση και τώρα χρόνια ολόκληρα δεν έχουν ε, κάνει τίποτα. Δεν αρκούν αυτά. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ βοηθήστε τον κόσμο αυτόν. Εγώ ευτυχώ, δεν είμαι ανάπηρος. Είναι όμως πραγματικά γελίο αυτό για όσους είναι ανάπηροι το γεγονό ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν, δεν μπορούν να ταξιδέψουν καν στο χωριό του χωρίς να έχουν προβλήματα προσβασιμότητας. Είναι πραγματικά λυπηρό και φρικτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Εξ όσων καταλαβαίνουμε, εμείς ως Επιτροπή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα τυπικά και επίσημα. Εμείς μαζί με εσά και μαζί με άλλους εμπλεκόμενους φορείς ασφαλώς μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οδηγία ίσης ε, μεταχείρισης, το οποίο και ασφαλώς θα το κάνουμε. Θα λάβουμε υπόψη και τις ιδιαίτερες ανησυχίες που έχετε και εκφράσατε για την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ευρωπαϊκή πράξη, για την προσβασιμότητα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε. Και στη συνέχεια επαφίεται σε εμά να κάνουμε και λόμπι προς τα κρατημέλη για να φροντίσουμε ότι συμμορφώνονται απόλυτα με τις προδιαγραφές του ΟΗΕ και τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα, άνθρωπα, για τους άτομα με αναπηρία. Τι προτείνω λοιπόν, συνάδελφοι, αυτό ακριβώ να κάνουμε, να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση αυτή, αλλά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά, τυπικά και επίσημα, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτε. Ελπίζω να την. Προτείνω να την ε, κλείσουμε μετά τον διάλογο αυτό που έλαβε η χώρα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φανχέλντερ, για την συμβολή σα και την συμμετοχή σα, σα ευχαριστώ για το γεγονό ότι καταλαβαίνετε ότι ω θεσμικό όργανο παρακολουθούμε το θέμα. Συνάδελφοι, συμφωνείτε να κλείσει η αναφορά αυτή με τη δέσμευση της ε, συνεχιζόμενης παρακολούθησης ε, του θέματο. Πολύ ωραία. Και περνάμε τώρα στην αναφορά 1294. Sorry. Mrs. Kuneva. Δεν σα είδα. Ναι, ναι, Ο λόγο είναι για εσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε που τελευταία στιγμή πανεύω. Νομίζω δεν, δεν φέρει τίποτα κανένα όφελο σε αυτό να κλείσω με την καταγγελία αυτή και το θέμα. Και αφού υπευθύνομαι σε εμά, πρέπει να κάνουμε κάποιε κινήσει, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε κάποιε κινήσει, προτάσει, συμμετοχέ, σε τροπολογίε για ώστε να βοηθήσουμε να εξελίξει αυτό. Γιατί πραγματικά είναι θέμα. Εγώ πριν να έρθω στο Κοινοβούλιο, συμμετείχα στο Σύλλογο των Τυφλών στο Παρίσι και ξέρω ακριβώ τα προβλήματα. Έχω παρακολουθήσει και εκπαίδευση σκύλων, έχω φίλου που έχουν ε, σκυλιά και ξέρω πόσο είναι ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση παντού γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε ραντεβού πουθενά. Έπρεπε να, να κατόμαστε όρθιοι στι πλατείε και στου δρόμου ή να μπούμε σε ένα σπίτι, το οποίο συνήθω δύσκολο γινόταν, για να έχουμε το ραντεβού και να συζητάμε. Αυτό είναι άνθρωποι τυφλοί. Έτσι. Και έρχονται από διάφορε περιοχέ κάπου για να κάνουν μια δουλειά, για να μπορούν να έχουν συνένεση και να μπορούν να συζητήσουν. Χρειάζονται στήριξη και από εμά. Δεν μπορούμε να μην έχουμε τη φωνή και να το στηρίξουμε. Βέβαια, εγώ συμφωνώ ότι σε κάποιο περιβάλλον μπορεί να προκαλούν αλλεργία και προβλήματα σε άσμα οι τρίχες των ζώων, αλλά εκτό από αυτό, με λίγο περισσότερη παιδεία στη κοινωνία, μπορούμε τα πράγματα να είναι πολύ πιο ομαλά και ωφέλιμα για όλους μας. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, then we do the following. Ε, ας κάνουμε λοιπόν το εξή. Μια και η κυρία Κούνεβα επιθυμεί να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, ας παραμείνει λοιπόν ανοιχτή. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως ανέφερα και προηγουμένως. Εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη αναφορά. Όχι, όχι στο σημείο αυτό πρέπει να συνεχίσουμε γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο μας και με το προηγούμενο εργαστήριο. Ή 11.40. Όχι. Η 12.94 διευθύνει η Πρόεδρος για την αχρωματοψία, ζητήματα αχρωματοψίας. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν και γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπάμαι που ξαναπαίρνω το λόγο. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που τέθηκε για τα άτομα που πάσχουν από δαλτονισμό και νομίζω ότι αυτό το θέμα της προσβασιμότητας που ελήφθη υπόψη και στα πλαίσια του European Accessibility Act που είναι υποσυζήτηση από Συμβούλιο και Κοινοβουλίο στο παράρτημα του εγγράφου προσθέτουμε μία σειρά λειτουργικών απαιτήσεων που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων που υποφέρουν από χρωματοψία. Υπάρχει και μια εντολή ε, που ουσιαστικά δόθηκε το 2005 στους οργανισμούς τυποποίησης και υιοθετήθηκε και ουσιαστικά αφορά αυτό το θέμα. Για να επανέλθω λοιπόν τώρα στι σημερινέ συζητήσει, ελπίζω ότι θα υπάρχει πρόοδος ε, χάρη στην υιοθέτηση της πράξη προσβασιμότητα που εξακολουθεί να είναι υπό διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Επιτέρα. Ευχαριστώ. Εγώ θα πρότεινα να κλείσει αυτή, αυτή η αναφορά. Αυτό το θέμα έχει να κάνει με την αχρωματοψία και ξέρετε ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν κάποια σήμανση λειτουργούν βάση ποσοστού. Παραδείγματο χάρη έχουμε διάφορες συσκευέ, ε, όπως ε, παραδείγματο χάρη ηλεκτρικέ συσκευέ ε, στην κουζίνα, όπου δεν έχουμε διαφορετικά χρώματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί λοιπόν να βάλει κάποιος μια σήμανση στις συσκευές που να δηλώνει το χάρη ότι έχει πάυσει η λειτουργία τους. Εγώ δεν πάσχω από αχρωματοψία, όμως μπορώ να καταλάβω πότε σταματάει ένα πλυντήριο ή πότε σταματά μια άλλη συσκευή και πώς η ενέργεια καταναλώνει. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και προτείνω να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, γνωρίζει αυτά τα θέματα και προσπαθεί να τα επιλύσει μέσω της νομοθεσίας και μέσω των διάφορων προτύπων στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να στείλουμε την απάντηση της Κομισιόν στον αναφέροντα και κατόπιν να κλείσουμε την αναφορά όπως είπε η κυρία Πιτέρα. Μπορώ να το πράξω αυτό, συμφωνείτε, μάλιστα. Ευχαριστώ. Ωραία. Περνάμε τώρα, κάπως ε, γρήγορα κινούμαστε. Το ξέρω, αλλά πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί γιατί καθυστερήσαμε το πρωί. Η επόμενη αναφορά είναι η 1123 και αφορά τη μία αναγνώριση της αυστριακής νοηματικής γλώσσας ως πρώτης γλώσσας ε, των υπήκων της Αυστρίας που είναι κοφή. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον αναφέροντα, τον Φραντς Ντότερ, στην Επιτροπή μας σήμερα το πρωί και να σας δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ που αναφέρεστε στο θέμα αυτό. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον ε, μπορεί να εκπληρωθεί η επιθυμία που έχω, γιατί εγώ τι θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Αναφορών συγκεκριμένα, να ε, φτύνει έκκληση προς την Αυστριακή κυβέρνηση για να σταματήσει η άδικη μεταχείριση των κοφών στη χώρα μας. Δεν πρόκειται να συζητήσω τα θέματα των κοφών γιατί ο κύριος Κόουσα, η κυρία Στέβενς που είναι το πέρα είναι εκπρόσωποι των κοφών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα ωστόσο να αναφέρω γιατί θα πρέπει να απευθυνθεί έκκληση προς την Αυστρία. Καταρχάς, σε θέματα γλώσσα. η Αυστρία δεν είναι και τόσο πίσω. Η Αυστρία έχει καλούς, καλή νομοθεσία για τις γλωσσικέ μειονότητες, τι αυτόχθονες γλωσσικέ μειονότητε σε ό,τι αφορά την προφορικό λόγο. Και επίσης έχει και καλή νομοθεσία για τα παιδιά των μεταναστών η Αυστρία για να υπάρχει σωστή ενσωμάτωση. Άρα οι γλώσσες των ε, μεταναστών επίσης λαμβάνονται υπόψη από την διοίκηση. Παρ' όλα αυτά, η Αυστρία δεν δίνει τα ίδια δικαιώματα προς τους κοφούς. Και δεν εξανίσταμε και ζητώ υποστήριξη και έκκληση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη απλή άρνηση. Είναι η άδικη μεταχείριση των κοφών που με αγανακτεί. Η άδικη μεταχείριση των κοφών όταν ζητούν να αναγνωριστούν τα δικαιώματά του. Και εδώ να εξηγήσω το εξή. Καταρχά, υπάρχει συνταγματική ρύθμιση η οποία την προβλέπει σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συνθήκες το Αυστριακό Κοινοβούλιο δεν ξέρουμε κατά πόσον οι διεθνείς συνθήκες αυτές πραγματικά μπορούν να μεταφερθούν σε αυστριακό δίκαιο. Αυτό είναι ένα πρακτικό πολιτικό εργαλείο εκ πρώτης όψεως. Αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνεται όσο η Αυστρία δεν έχει αποφανθεί και δεν υπάρχει εθνικό δίκαιο, δεν έχει καμία σημασία η διεθνή συνθήκη, το διεθνές δίκαιο. Αυτή η πολιτική της ε, Αυστρίας, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έχει αποτεχθεί δηλαδή η Αυστρία τη διεθνή συνθήκη. Υπάρχει όμως από το Κοινοβούλιο μια νομική επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τη σύμβαση, τη συνθήκη του ΟΗΕ. Αυτό τι σημαίνει ότι κανείς, κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να, να επικαλεστεί τη σύμβαση αυτή. Άρα, έχει αποδεχτεί μεν η Αυστρία τη σύμβαση του ΟΗΕ, αλλά στην πράξη, στην καθημερινή δουλειά, δεν χρησιμοποιείται. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες χώρες. Αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν ε, συνάδει με το γράμμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και με τις ευρωπαϊκές αξίες. Ούτε καν με τις αυστριακές. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω. Στις ε, διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για, την, για τα δικαιώματα των αναπήρων βλέπουμε μια πρακτική της κυβέρνησης, την εξή. Θέλουν πραγματικά να καταλύσουν αυτές τις διαδικασίες μέσω ψευδών κοινοποιήσεων, για παράδειγμα. Αν ένα κοφός απευθυνθεί προς μια υπηρεσία για να κάνει μια αίτηση, ιδιαίτερα στην νοηματική, για την νοηματική στην εκπαίδευση, για παράδειγμα. Τότε η κυβέρνηση ξέρει και έχει υπόψη τη ότι χρειάζεται μια σωστή κοινοποίηση για να μπορεί κανεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο για θέματα συνταγματικά, για παράδειγμα. Αλλά πολύ απλά δεν παίρνει ο πολίτης τη σωστή κοινοποίηση. Άρα ουσιαστικά πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η ψευδής ε, κοινοποίηση. Και η τρίτη στρατηγική που με εξοργίζει είναι ότι η Αυστρία παρουσιάζει επιχειρήματα τα οποία τι λένε. Όταν ρωτάει κανείς ε, γιατί δεν δίνετε δικαιώματα στους κοφούς, απαντάνε, α, κάνουμε τόσα πολλά επιπλέον και παραπάνω από αυτά που ορίζει η νομοθεσία. Αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Με ξεπερνάει. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάρκετ, την πλευρά τη Κομισιόν. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξή. Η Κομισιόν ε, προωθεί τη χρήση της νοηματικής για τους κοφούς στο πλαίσιο της πυκλομορφίας των γλωσσών στην Ευρώπη, αλλά και στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των ατομών με αναπηρία. Αλλά ως κανόνας, όπως ξέρετε, η Ένωση μπορεί να δράσει εντός των αρμοδιοτήτων που της δίνει συνθήκη. Και στην περίπτωση αυτή, τα θέματα που τέθηκαν είναι αποκλειστικές αρμοδιότητας των κρατών μελών. Δηλαδή πρόκειται για την οργάνωση των ε, εκπαιδευτικών συστημάτων. Η Κομισιόν επομένω δεν μπορεί να διερευνήσει νομικά αυτά τα θέματα. Ακόμη και αν ε, η αρχή της ε, μη διάκρισης έχει εγγραφεί στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η διάταξη της Χάρτας δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν εφαρμόζεται εδώ Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης, η Κομισιόν δεν μπορεί να διερευνήσει νομικά τα θέματα μη συμμόρφωση με τις διεθνείς ε, υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες πηγές πέραν των Ευρωπαϊκών Συνδικών όπω ε, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρωπινά Δικαιώματα ή τι συμβάσει του ΙΕ. Δεν μπορεί η Κομισιόν να, ε, να διερευνήσει τέτοιες πτυχές, ούτε μπορεί να σχολιάσει για το αν γίνεται σεβαστό το Αυστριακό Σύνταγμα ή αν έχουν θεσπιστεί εθνικές αρχές που συνάδουν με τις συνταγματικές διευθετήσεις ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό το θέμα όμως ε, δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό. Φυσικά πρέπει αυτά τα θέματα καταρχήν να λυθούν σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους, αν θέλουν να παρέμβουν, κυρία Τανόκα. Ευχαριστώ. Αυτό που ακούσαμε μόλις από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν είναι μια πρότυπη απάντηση, μια τυπική απάντηση ότι Έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα λοιπόν του κράτου μέλου. Όμως, τι ζητά ο αναφέρον. Μας ζητά να απευθυνθούμε στις αρχές της Αυστρία. Και είναι δική μας αρμοδιότητα να το κάνουμε αυτό. Και θέλω να υποστηρίξω το αίτημά του. Ναι, πρέπει να κάνουμε μια παραπομπή στη χάρτα. Διαφορετικά, γιατί αποτελεί μέρος των συνδικών η χάρτα. Διαφορετικά θα ήταν απλώ ένα κομμάτι χαρτί. Νομίζω ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στι αυστριακές αρχές και να τους υπενθυμίσουμε την υποχρέωσή του Ναι, είναι αρμοδιότητα κρατική, αλλά το κράτος πρέπει να λάβει υπόψη και τα ευρωπαϊκά έγγραφα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Κώσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, ακόμη και αν δεν είμαι μέλος της Επίτροπος Αναφορών, θα είμαι σύντομος. Όμως, όπως και να έχει, αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι ότι η αναφορά που παρουσιάστηκε έχει να κάνει με την κατάσταση στην Αυστρία. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν απαντάται μόνο στην Αυστρία. Είναι κάτι που συμβαίνει στην πράξη και πλήττει τους κοφούς σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια καταγγελία που έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά όπως ε, είπε και ο Αναφέρον, ε, η διάκριση αυτή δεν γίνεται μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά σε όλους ε, τους τομείς που αφορούν τη ζωή των κοφών παιδιών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει και την κατάσταση αυτή, η ίδια αναφορά γίνεται και στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και εγώ νομίζω γι' αυτό είναι ευθύνη της Επιτροπής Αναφορών να απευθυνθεί στην Αυστριακή κυβέρνηση για να τη ρωτήσει τι γνωμοδοτεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα που εντοπίζεται αποκλειστικά στην Αυστρία, εγώ όμως πιστεύω ότι ίσως οι συντονιστές της Επιτροπής Αναφορών θα μπορούσαν να εξετάσουν το να εκπονηθεί μια έκθεση για την πρόσβαση των κοφών παιδιών στις διάφορες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες εκπαίδευσης. Και για να κλείσω, θέλω να πω ότι εδώ συζητάμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Τα κοφά παιδιά λόγω της αναπηρίας τους μπορεί να θεωρηθούν και ότι αποτελούν και μια γλωσσική μειονότητα. Η δική τους μητρική γλώσσα είναι η νοηματική, στη συγκεκριμένη περίπτωση η αυστριακή νοηματική, στη Σουηδία η σουηδική νοηματική γλώσσα. Για μας η νοηματική γλώσσα είναι η πρώτη μας γλώσσα και εδώ μιλάμε για περιορισμό στην άσκηση των γλωσσικών δικαιωμάτων. Επομένως, θα ήθελα να ζητήσω να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά και να απαντήσει η αυστριακή κυβέρνηση στο τι συμβαίνει. Και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι θα ήταν καλό να εκπονηθεί και μία έκθεση για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ Γιάρ. Ναι, φυσικά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε βράχη πρόθεσμα και πρόθεσμα Βράχη πρόθεσμα όμως πρέπει να αντιπιστώσουμε ότι αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό λοιπόν καλό καταπηγόντως τον αναφέροντα να απευθυνθεί και στην ε, Επιτροπή Αναφορών στην Αυστρία. Εκεί μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα το θέμα. Τις άλλες ε, απαντήσεις προς την Πρόεδρο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. να ρωτήσουμε όλα τα κράτη-μέλη κατά πόσον υπάρχει μια ε, ξεχωριστή επιτροπή, αρμόδια επιτροπή που ελέγχει τα πράγματα στις χώρες. Γιατί υπάρχει και θέμα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. Γιατί φυσικά είναι θέμα διακριτικής μεταχείρισης, αλλά αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη. Σίγουρα λοιπόν ο αναφέροντας να μην αμελήσει να απευθυνθεί στην Αυστριακή Επιτροπή αναφορών να υποβάλει τέτοια αξίωση και αναφορά για να συζητηθεί επιτόπου το θέμα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ανέφερε και η Επιτροπή, από νομικής πλευράς δεν μπορεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο η Επιτροπή Αναφορών για αυτό το θέμα, επειδή είναι αναφορά που σχετίζεται με εθνικές αρμοδιότητες εμπίπτει στις εθνικές αρμοδιότητες. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι μερικές φορές μπορούμε να δράσουμε κατά τρόπο που να είναι ευεργετικός για τους αναφέροντες, αν και από νομικής πλευράς δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Δηλαδή, αρκετές φορές είδαμε ότι βοηθά μία επιστολή προς τις εθνικές αρχές. Θα πρότεινα λοιπόν να αποστείλουμε μία επιστολή στις αυστριακές αρχές, όπου να αναφερόμαστε στις πρακτικές αυτές διακρίσεων κατά των φυσικών αυτών προσώπων, να αναφερθούμε στην πράξη προσβασιμότητας και το γεγονός ότι εμείς εποπτεύουμε αυτό το πλαίσιο. Να το καταστήσουμε δηλαδή απόλυτα σαφές. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Όμως θα πρέπει να κλείσουμε την αναφορά κύριε Ντότερ, δεν μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα για σας. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να αποτανθείτε στην Αυστριακή Επιτροπή Αναφορών, γιατί εμπίπτει σε, στις εθνικές αρμοδιότητες. Συνάδελφοι, η κυρία Άουκεν ζήτησε το λόγο. Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, γιατί πρόκειται για θέμα συναπόφασης όταν μιλάμε για θέματα νικής υφής. Όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα ε, θέματα που προκαλούν ε, διακρίσεις σε σχέση και με ενδεχόμενα ένδικα μέσα. Έχουμε ασχοληθεί με ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία εγγράφονται στις συνθήκες μας. Γι' αυτό θα ήθελα περιμένουμε την απάντηση από τις Αυστριακές Αρχές. Συμφωνώ, μαρκρίτ αλλά καταρχήν ε, εγώ ε, είμαι με, την πλευρά, είμαι στην πλευρά του αναφέροντος και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζεις πολύ καλά ε, εσύ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο δέχεστε αυτό που πρότεινα. Δέχομαι την ε, ιδέα της επιστολής. Θα δεχτώ τη σύσταση του Γερμανού Ευρωβουλευτή και θα ε, αποτανθώ στην Αυστριακή Επιτροπή αντιμετώπισης των αναπηρεών, δηλαδή στην Αυστριακή Επιτροπή Αναφορών. Χρειαζόμαστε αυτή την επιστολή γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη βούληση από πλευράς Αυστριακών αρχών. αλλά τα ένδικα μέσα διαρκούν τόσο πολύ, η προσφυγή στα δικαστήρια δηλαδή, ώστε ε, μέχρι να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά που είναι τώρα μαθητές ε, θα έχουν γίνει ενήλικες. Είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία. Λοιπόν, Ε, ο αναφέρον θα αναφερθεί στην Επιτροπή Αναφορών της Αυστρίας και εμεί θα αποστείλουμε επιστολή στις Αυστριακές Αρχές και κλείνω την αναφορά. Ωραία, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι όταν όλοι είναι ικανοποιημένοι και στρεφόμαστε στην επόμενη αναφορά 240 σε σχέση με τελωνιακές ατέλειες από εισαγωγικούς δασμούς που σχετίζονται με την εκπαιδευτική, επιστημονική και μορφωτική πραγωγή των ε, ατόμων με αναπηρία. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν, ίσως μας παρακολουθεί μέσω ε, διαδικτύου και δίνω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Ματίας Μπιόργ Λαντ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μία περίπτωση όπου ο κύριος Γκαβρίλα ήρθε σε άμεση επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς ήρθαμε σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές και συμφωνήσαμε ότι ο εθνικός νόμος καλύπτει μόνο εν μέρη τέτοια ζητήματα όπως ε, τον κανονισμό του 2009 για τους τελωνιακούς δασμούς και τις ατέλειες. Και θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εφαρμογή αυτού του κανονισμού, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο δυσχερές λόγω των ε, ανεπαρκειών. Ε, ε του άρθρου 257 των συνθήκων έγινε προσφυγή επί παραλήψη. Ο κύριος Γκαβρίλα διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το ζήτημα άμεσα, σε σχέση δηλαδή με τους τελωνιακούς δασμούς δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού. Μετά από τις επαφές μας, οι Ρουμανικές αρχές θα αναστείλουν αυτή την νομοθεσία, θα την ανακαλέσουν και γι' αυτό θα κλείσουμε εμείς το ζήτημα αυτό γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει πλήρης εφαρμογή του κανονισμού. Γράψαμε στον κύριο Γκαβρίλα, αλλά μας ξαναέγραψε ότι κατά την άποψή του ε, το περιεχόμενο της ανάκλησης αυτής η ανάκληση αυτή αφορά ε, και ένα ε, νέο κανονιστικό πλαίσιο 105 κάθετος 16. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε αυτό το ζήτημα γιατί τώρα μελετούμε τα νέα στοιχεία που λάβαμε στις 28 Οκτωβρίου. Αλλά από πρώτη ματιά η ανάκληση αυτή αφορά τον ΦΠΑ και όχι ε, την εξάλληψη τελωνιακών ε, δασμών. Άρα μιλάμε μόνο για ΦΠΑ και όχι γενικά για τελωνιακές ατέλειες. Αυτή είναι η πρίμα φάση ε, αποτίμηση της κατάστασης. Άρα θα πρέπει να μελετήσουμε εις βάθος το θέμα πριν κλείσουμε το ζήτημα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχουν τα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Τανόκα. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε, να αφήσουμε μάλλον την αναφορά ανοιχτή και να περιμένουμε τη νέα νομοθεσία. Το θέμα είναι σχετικά απλό. Σύμφωνα απόλυτα δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς, άρα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά μέχρι την απόλυτη διασάφηση του ζητήματος. Ζητούμε από την Επιτροπή να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση και να μας γράψετε όταν έχετε νεότερα. Εντάξει, ωραία. Το επόμενο θέμα είναι η αναφορά 924 του Νταν Πέσκοτ εξ ονόματος του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών σε σχέση με την πρόσβαση των ε, τυφλών ε, σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα και επίσης αναφορά 9-6-4 για τους δυσλεκτικούς, για τα άτομα με δυσλεξία και άλλες αναπηρίες και την πρόσβασή του στα βιβλία. Δίνω το λόγο στον David για 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι η εξαιρετική έρευνα και μελέτη που έγινε για την σύμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της πολιτικής. Η συνθήκη του Μαρακές, λοιπόν, ήταν εξαιρετική και δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η μελέτη ε, για την συνθήκη του Μαρακές χωρίς τα, την εργασία της Επιτροπής ε, Αναφορών. Να το έχουμε αυτό υπόψη. υπόψη. Και τώρα λοιπόν έχει έρθει η στιγμή να, κάνουμε και, να καλύψουμε και την τελευταία απόσταση, το τελικό κομμάτι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή χωρί νομικά προβλήματα, χωρί νομικέ επιβεβαιότητε, χωρί εμπόδια και ναι με 25 έω 30 χώρε έχουν επικυρώσει τη συνθήκη, αλλά η συνθήκη της του ξέρετε, δεν πρόκειται να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο, εκτός κι αν επικυρεώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εδώ ε, μιλάμε για τεράστιο όγκο ψηφιοποιημένων βιβλίων και έντυπων προϊόντων. Και ιδιαίτερα τώρα με το εκλογικό αποτέλεσμα που ακούσαμε σήμερα το πρωί από τη ΣΥΠΑ, πολύ φοβάμαι ότι επικρατεί μεγάλη ανησυχία γιατί υπήρχαν ελπίδες για επικύρωση από πλευρά των ΙΠΑ αλλά τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει γιατί οι ΙΠΑ ασφαλώς αποτελούν την άλλη μεγάλη δύναμη σε ό,τι αφορά τα ψηφιοποιημένα έντυπα προϊόντα. Άρα είναι επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες αυτά τα βιβλία. Και πιο πολλές γλώσσες είναι εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ζητούμε καταπηγόντως επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω νομοθεσίας. Χαιρόμαστε με την πρόσφατη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οδηγία και κανονισμό. Αποτελεί μια γενικότερη αποτύπωση των γενικότερων στόχων και αναγκών για τα άτομα ε, που έχουν πρόβλημα όραση και εκπροσωπώνται παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών και την Διεθνή ε, Ένωση Τυφλών. Θέλουμε λοιπόν να εγκριθούν αυτά από το Συμβούλιο χωρίς να προσθεθούν νομικά εμπόδια. Συζητιούνται κάποια νομικά εμπόδια από κάποιες χώρες για διάφορα στοιχεία που τους ανησυχούν. Ένα από αυτά είναι η εμπορική διαθεσιμότητα. Αυτό τι σημαίνει ότι αν μπορεί κανείς να αγοράσει ένα βιβλίο οπουδήποτε στον κόσμο, δεν μπορεί ουσιαστικά να το μοιραστεί. Αυτό θέλει να προτείνουν κάποιους αυτό θεωρώ ότι αποτελεί διακριτική μεταχείριση. Γιατί ω ε, άτομο που δεν έχω αναπηρία μπορώ να πάω να αγοράσω ένα βιβλίο και να το χρησιμοποιήσω όπως θέλω. Θεωρώ ότι αυτό θα δημιουργούσε μεγάλη νομική αβεβαιότητα. Θα σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνονται τεράστιες ε, έρευνε και αναζητήσει και ότι δεν θα είχαν συμφέρον οι εταιρείε να δημοσιεύσουν τα βιβλία αυτά σε ε, ψηφιοποιημένη μορφή. Γιατί αυτό αποτελεί και τον στόχο της συνθήκης του Μαρακές ουσιαστικά. Γιατί διαπιστώνουμε ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση μόνο σε 1% των συνολικών αντίπων προϊόντων. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να περιπλέξει περιττώρο την κατάσταση σε ό,τι αφορά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα διοικητικά εμπόδια και ακόμα και το κοινοβούλιο. Αυτό αναφέρεται και στη μελέτη του Τμήματο πολιτικής ανάλυσης. Θα μπορούσε να εξετάσει κάποιες πιο τεχνικές ε, διαστάσεις που θα μπορούσαν να κάνουν την συνθήκη πιο αποτελεσματική. Στα ακουστικά να επεκταθούν οι διατάξεις, τις συνθήκες και να εφαρμοστεί αυτό και για άλλα άτομα με άλλα αναπηρία. Τι ζητούμε λοιπόν. Ζητάμε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα καταρτήσει γνωμοδότηση για τη νέα οδηγία και τον νέο κανονισμό. Δεν ξέρω, γιατί αποφασίσει να γίνει σχετική γνωμοδότηση, μάλιστα, καταφατική απάντηση, να συνεχίσει να επιδεικνύει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί και να προσπαθεί να προσπαθήσει να συνενώσει την Επιτροπή, του Σύμβουλου και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων προκειμένου να υπάρχει μια γρήγορη ανάγνωση και α, πρόθεση του θέματος για να μπορέσει να ψηφιστεί αυτό την ερχόμενη άνοιξη στην Ολομέλεια. Να αναφέρω επίσης ότι το θέμα της αρμοδιότητας πλέον λίγο πολύ έχει επιληθεί με την γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελία, ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει νομική βάση να αντιταχθεί κανείς στην ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει ήδη μια νέα αναφορά που κατατέθηκε από την ενέργεια του τυφλών πριν από τρει-τέσσερι μήνες, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα θέματα επικύρωσης και εφαρμογής της συνθήκης. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τελευταία πρόταση, πρόεδρε. Να σας πω ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό, λοιπόν, συμμόρφωσης. Έναν μηχανισμό υποβολής ενστάσεων, ένα σχέδιο δράσης από προβλημάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα εφαρμοστεί η συνθήκη του Μαρακές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τον ρόλο που διαδραματίσατε και να δώσω τον λόγο στον συνάδελφό μου από την οργάνωση των ατόμων με τη δυσλεξία. Έχετε το λόγο, λέει η Πρόεδρος. Καλημέρα σας, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εκμορφωπώ τον κύριο Κάλμαρ, τον Αυστριακό Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δυσλεξίας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι, ότι υποστηρίζουμε την κύρωση της συνθήκες ε, του Μαρακές ε, για ε, όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δυσλεξία ή άλλες μαθησίκες δυσκολίες και φυσικά αναφέρεται ότι είναι σημαντική για την πρόσβαση στη ψυχαγωγή και στον πολιτισμό. Βεβαίως είναι ε, σημαντική και η Ρωσία αυτή τη σύμβαση, αλλά είναι και σημαντική η πρόσβαση ε, των παιδιών με αναπηρία σε βιβλία για να μπορούν ε, να φτάσουν σε επίπεδα τυχείων που δεν έχουν σήμερα και είναι και σημαντικό και για τη διαβίου κατάρτιση Συμφωνώ όμως είπε ο συνάδελφος Ντέιβιτ ε, ε, και πρέπει να μπορούν ε, οι άνθρωποι να περιέχουν να διαβάζουν βιβλία που πολλές φορές δημοσιεύονται και σε άλλες χώρες, σε άλλες γλώσσες και θα πρέπει να μοιράζονται τα κείμενα και να υπάρχει και ένας καλός βαθμός προσβασιμότητας στα βιβλία αυτά. Επίσης είναι και θέμα πρόσβαση στην ηθαγένεια. Όταν ε, δεν έχουμε πρόσβαση στα βιβλία, πώς μπορούμε να είμαστε πολίτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Πολλοί πολίτες ε, δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Έτσι λοιπόν για τα άτομα που έχουν συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες ή πολύ σοβαρέ δυσκολίες ε, που τους εμποδίζουν να διαβάσουν καθόλου ή άλλες ε, πιο ε, όχι τόσο σοβαρές δυσκολίες. Η πρόσβαση στα βιβλία είναι απαραίτητη για κάποιους, είναι πολύ χρήσιμη για άλλους και είναι κάτι πρακτικό και χρήσιμο για όλους. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών προκειμένου στα κράτη-μέλη να προχωρήσει η κύρωση της σύμβασης του Μαρακές και έτσι ώστε να μπορούν να βοηθηθούν και οι τυφλοί αλλά και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ανάγνωσης εντύπων που είναι print disabled λέει ο μιλτής. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Το Τόμας την είναι Κομισιόν. το λόγο. Καλημέρα σας. Καταρχήν, θα θέλαμε να δράξουμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τερμισμόντες ε, για την παρουσίαση σήμερα το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που αναφέρονται σε αυτήν την αφορά, θέλουμε και εμείς να αναφέρουμε ότι τελικά υπάρχει μια κίνηση παρατηρείται προς το θέμα της κύρωσης ε, και μετά τις 8 Σεπτεμβρίου τώρα αναμένουμε την γνωμοδότηση του δικαστηρίου πολύ σύντομα. Έτσι ώστε το θέμα της αποκλειστικής ή της μικτής αρμοδιότητας να επιληθεί εν τέλει και να είμαστε σε θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθούμε γρήγορα με την κύρωση της συνθήκης. Επίσης, ακούσαμε με χαρά ότι οι προτάσεις μας για την εφαρμογή της ε, συνθήκης, της οδηγίας και του κανονισμού. Απαντώνται με πολύ θετικό τρόπο από τους αναφέροντες. Υιοθετήσαμε αυτή την πρόταση στα μέσα Σεπτεμβρίου και τώρα έχουμε τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Ξεκίνησαν τον Οκτώβριο και έχουμε και την πρώτη ακρόαση, την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Γιούρη, στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα νομίζω. Και μπορούμε να παρευρεθούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις φυσικά και να δούμε την σύντομη ολοκληρωσή τους. Ό,τι αφορά το θέμα άλλων αναπηριών, ένα θέμα που θυχτήκε και από τους δύο αναφέροντες, θέλω να τονίσω ότι στην οδηγία, στο άρθρο 7, έχουμε συμπεριλάβει μια έκθεση που θα πρέπει να ελοπιθεί εντός δύο ετών μετά τη θέση εφαρμογή της οδηγίας και που θα επικεντρώνεται στην κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά άλλες αναπηρίες και αυτό είναι ε, ουσιαστικά υποχρέωσή μας ε, στα πλαίσια της αρχής της καλύτερης νομοθεσίας. Αυτά προς το παρόν θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στους αδέλφους Μάρκαρτ. Νομίζω ότι θα πρέπει να γιορτάσουμε. Είχαμε τώρα αυτή την αναφορά και το θέμα στην ημερήσια διάταξη για τόσο πολύ καιρό. Και ενίοτε ένα, γιορτάζαμε, μετά σημειώναμε ήττα. Και νομίζω ότι ήταν ε, πραγματικά σοκαριστικό για να δούμε ότι υπήρχαν διάφορα συμφέροντα που ήθελαν να μπλοκάρουν ε, ε, αυτούς τους ανθρώπους, τους τυφλούς και τα προβλήματα, τα προβλήματα να έχουν πρόσβαση στα βιβλία. Και εδώ μας υπενθύμησαν ότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και η Ευρώπη έχει το κλειδί. Έχουμε πάρα πολλές γλώσσες Επομένως, εδώ έχουμε ένα ρόλο κλειδί να διαδραματίσουμε. Εκτιμώ ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα και ελπίζω ότι θα είμαι και εγώ σε ηγετική θέση στις διαπραγματεύσεις. Και ελπίζω ότι θα έχω πάρα πολύ καλές και ενθουσιώδεις συνεισφορές. Γιατί κάποιοι εξημών ε, έχετε δώσει αυτή τη μάχη ήδη τα τελευταία 5-6 χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την αναφορά. Thank really Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πραγματικά είναι πολύ καλή ημέρα για την Επιτροπή Αναφορών. Καταρχάς είχαμε το εργαστήριο σήμερα το πρωί και τώρα. Αυτή η αναφορά, όπω ε, όπως είπατε, μας απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πάει καλά. Πέτερ. Ναι, υποστηρίζουμε ασφαλώς ε, την θέση αυτή και νομίζω ότι όπως είπε η Μάρκαρετ ελπίζουμε να πετύχουμε και το τελικό αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε ως Επιτροπή Αναφορών. Θα πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμόζονται τα όσα αποφασίζονται. Καλή ημέρα. Αλλά, Μάργαρετ, να διανύσουμε για αυτήν την τελική απόσταση για να μπορέσουμε πραγματικά να γιορτάσουμε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κλείσουμε με το θέμα αυτό. Συμφωνεί απόλυτα και συμφωνούν απόλυτα και οι αναφέροντες. Και όπως ξέρουμε, για το θέμα αυτό αρμόδια είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θα χρειαστεί και η έγκριση του Κοινοβουλίου για την επικύρωση. Μαξ Άντερσον είναι ο υπεύθυνο και για τις τρεις, τα τρία θέματα που έχουν να κάνουν με τις αντικτυμαρασικές. Είναι πράσινος, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός και πολύ ευγενή Και εξ ονόματος της Επιτροπής αυτής Υπάρχει ήδη μια απόφαση ότι θα γνωμοδοτήσουμε προς την Γιούρη, προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η Μάργαρετ Άουκεν θα αναλάβει το έργο αυτό και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Τυπικά αυτά. Τώρα, στο πνεύμα της 0924 ε, θα συνεχιστεί από την καινούργια αναφορά που ήδη αναφέρθηκε και έχει ήδη κατατεθεί σε ό,τι αφορά την ε, ταχεία εφαρμογή και επικύρωση, συγγνώμη, της συνθήκης του Μαρακές. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, να κλείσουμε την 0924, η επόμενη ιδέα αναφορά, η οποία είναι πιο ενημερωμένη, πιο σύγχρονη. Θα παραμένει ανοιχτή μέχρι ότου να ολοκληρωθεί με τον επιτυχή τρόπο. Ναι, ναι, ναι μισό λεπτό. Νομίζω ότι η 0924 εξυπηρέτησε το σκοπό της και όπως είπε και η Μάρκαρετ μπορούμε να γιορτάσουμε σήμερα. Για άλλη τώρα η αναφορά. Η 964 να ζητήσω από τον αναφέροντα να καταθέσει καινούργια αναφορά εφόσον το επιθυμεί. Και να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε και την 964 που επίσης είναι παροχημένη. Το θέμα όμως ασφαλώς παραμένει ανοιχτό και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση και τα δύο νομοθετικά αρχεία που έχουν να κάνουν με τη συνθήκη του Μαρακέσου. Συμφωνείτε συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Για να δω. Άλλη μία αναφορά έχω πριν το μεσημέρι. Για ένα μισή λεπτό θα σας το λέω. Το πρόβλημα στην όλη αυτή τη διαδικασία δεν ήταν ε, το Κοινοβούλιο, αλλά κάποια κρατημέλη στο Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και νομίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να βοηθήσει και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων προκειμένου τα όσα συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο να παρακολουθούν πιο στενά γιατί από τι ομάδε εργασία του Συμβουλίου μας λένε ότι παντού υπάρχουν προβλήματα και είναι πολύ πιο διστακτική από ότι εδώ. Ζητώ λοιπόν από τους βουλευτές που είναι εδώ να έρθουν σε επαφή με τα κράτη-μέλη τους για να εξασφαλίσουν ότι όλα όσα θίξαμε και θήγηκε η Επιτροπή Αναφορών πραγματικά λαμβάνονται υπόψη στα Υπουργεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, και φυσικά αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Είναι... Ότι δηλαδή το Συμβούλιο είναι ένα διαφορετικό θεσμικό όργανο. Είμαστε από κοινού νομοθέτες, άρα πρέπει να συνεργαστούμε και από καιρού εις καιρών πρέπει να βγαίνουμε από τα χαρακόμματα και να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Αυτό είναι το θέμα ουσίας. Άρα να είσαστε ήσυχος. Η επόμενη αναφορά είναι η 845 εξ ονόματος των, ε, της Ρουμανικής και Γερμανικής Ένωσης Alsterdorf σε σχέση με τρεις ενώσεις ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στη Ρουμανία. Το λόγο έχει η Επιτροπή γιατί ο αναφέρον δεν είναι παρόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη λόγω ώρας. Θα ήθελα να σας πω απλώς, ε, όπως και στη γραπτή μας απάντηση, ότι πράγματι η κατάσταση στη Ρουμανία ως προς την αντιμετώπιση των ανθρώπων με αναπηρία ε, οδήγησε σε μία αντίγνωμη έκθεση του 2016 μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας 15-16. Άρα ε, εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ως και προς τη διάθεση πόρων και την ε, χρήση διαρθρωτικών πόρων μέσα στα πλαίσια και της Regio και της Amplua έτσι ώστε να μπορούν να ζουν σε ανοιχτές κοινότητες και να μην πάσχουν από ιδρυματισμό αυτά τα άτομα. Άρα είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στον τομέα αυτό. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, συνάδελφοι, ποιος θέλει το λόγο. Ο Πέτερ, από πλευράς πολιτικής ε, Σήμερα το πρωί είχαμε και το εργαστήριο. Μπορούμε να πούμε ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει αναγνωρίσει το θέμα αυτό ως πρόβλημα και σε ό,τι αφορά τη Σλοβακία το θέμα αυτό παρόμοιο ήταν και τότε. θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση. Ξέρουμε ότι δεν είναι απλά πράγματα. Το είδαμε και στην περίπτωση της Σλοβακίας. Υπάρχουν ε, όπου ενδεχομένως να υπάρχει βούληση, αλλά θα πρέπει να εξετάζει η Επιτροπή Αναφορών το θέμα. Να πούμε και στον αναφέροντα ότι γνωρίσαμε το πρόβλημα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε και με την διερευνητική αποστολή ήταν ε, σαφές, έγινε σαφές ότι το πώ θα καταλήξουμε από το α στο β είναι πάντα ένα πρόβλημα. Γιατί είναι σαφής ποιος είναι ο στόχος, αλλά πώς θα τον πετύχουμε, αυτό είναι το θέμα. Και θα ήθελα λοιπόν κάποια υποστήριξη προς την κατεύθυνση αυτή. Να παραμείνει λοιπόν ανοιχτή η αναφορά αυτή. Okay. I think Peter... Ωραία, νομίζω Πέτερ ότι κατέστησε τους συναδέλφους ε, ευτυχής. Αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά. Ναι, την αφήνουμε ανοιχτή και νομίζω ότι θα πρέπει να αποστείλουμε στις ρουμανικές αρχές μία ε, Πιστολή, ε, δυνάμει του, της Σύμβασης των Ηνωμένων ε, Εθνών και να τους ε, υπενθυμίσουμε τα καθήκοντά τους και να τους ενθαρρύνουμε να συμμορφωθούν. Ωραία. Τελειώσαμε με την πρωινή συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε στις 3. Γεια σας. Όχι αργότερα από τις 3. Γεια σας.